Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε συνάδελφοι στο νομισματικό διάλογο με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Μάριο Ντράγκη. Θέλω να τον καλωσορίσω και αυτόν. Είναι ο τέταρτος και τελευταίος νομισματικός διάλογος φέτος. Διεξάγεται αμέσως μετά <clears throat> μια σημαντική απόφαση στον τομέα το νομισματικό τον οποίο πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα πλαίσια μιας οικονομικής ανάκαμψης η οποία αυτή τη στιγμή αυξάνει την δυναμική της και νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται πιο σταθερή και με ευρύτερη βάση και ταυτόχρονα και εδώ ο κύριος Τράγκη θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία, βλέπουμε μια δυναμική τιμών, μια δυναμική τιμών η οποία δεν είναι ακόμα απόλυτα υποστηρίξιμη. Βλέπουμε μια δυναμική χαμηλών αμοιβών, χαμηλών μισθών και αυτό το είχαμε συζητήσει και στα πλαίσια του τελευταίου νομισματικού διαλόγου. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κυκλικοί διαρθρωτικοί λόγοι για τους οποίους, με τους οποίους εξηγείται το φαινόμενο αυτό των χαμηλών μισθών. Ο διάλογος αυτός ο νομισματικός λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντικός και οι αποφάσεις της Κεντρικής Τραπέζας είναι, η απόφαση είναι σημαντική να διατηρηθεί το quantitative easing, το QE, έτσι ώστε να πετύχει σε κάποια φάση τους στόχους της. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να έχουμε προβλήματα με τις καρέκλες. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Επανέρχεται ο κύριος Γκουαλτιέρη. Όπως γνωρίζει οι συντονιστές της ΕΚΟΝ έχουν επιλέξει κάποια επιμέρους θέματα όπως το ανισότητες και ελλείψεις ισορροπίας κατατομής, όπως επίσης και ε, η σταδιακή έξοδος από τα νομισματικά μέτρα, σε φάσεις έξοδος και τι σχέση έχει με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα. Υπήρξαν ορισμένες μελέτες εν το μεταξύ, κάποιες από αυτές μας λέγουν με πολύ πιστικό τρόπο το πώς οι ανισότητες αυτές αντικατοπτρίζουν κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά της ε, ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ή μάλλον της αρχιτεκτονικής του ευρώ. Εν πάση περιπτώσει αυτά είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι έχουν αρκετή σημασία. Σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά Πρόεδρε Ντάγη και σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές της Επιτροπής ε, Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, κυρίε και κύριοι. Χαίρομαι που βρίσκεμαι πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την τελευταία μου ακρόαση φέτο. Από την τελευταία μα συνάντηση, το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει λάβει σημαντικέ αποφάσει σχετικά με την αναπροσαρμογή των εργαλείων νομισματικής πολιτικής τη ε, πέρα από το τέλο αυτής της χρονιάς. Και γι' αυτό στι σημερινέ μου παρατηρήσει θα αναφερθώ πρώτα στις προβλέψεις ε, για την ε, οικονομία της ζώνης του ευρώ και την αναπροσαρμογή των μέτρων ε, νομισματικής πολιτικής μας. Κατόπιν, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής σας θα αναφερθώ στο Target 2 που στηρίζει τον, τη δημοσιονομική ολοκλήρωση και την εφαρμογή της νομισματικής μας πολιτικής που στη συνέχεια έχουν συνέπειες σχετικά με την ερμηνεία των ισοζυγίων Target. Η οικονομική διεύρυνση παραμένει σταθερή και ευρεία και στις διάφορες χώρες και στους διάφορους τομείς της ζώνης του ευρώ και στηρίζεται κυρίως από την ε, εγχώρια ζήτηση εγχώρια κατανάλωση. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ε, πρόβλεψη της Eurostat, η ανάπτυξη έχει συνεχιστεί στο τρίτο τρίμηνο της χρονιάς κατά 2,5% σε σχέση με πέρσι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 4,5 χρόνια συνεχούς ε, ανάπτυξης ε, κάθε τρίμηνο και τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η ορμή αυτή θα συνεχιστεί. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ επίσης ε, φαίνεται να υπάρχει σε όλες τις χώρες και τους τομείς. Και τα ποσοστά ανάπτυξης του ΑΕΠ, μάλλον η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά ανάπτυξης του ΑΕΠ έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1997. Έχουμε δηλαδή γενική προς τα πάνω σύγκληση. Η αγορά εργασίας ε, συνεχίζει να ωφελείται από την ανάκαμψη και οι βαθιές και επώδυνες ε, απώλειες ε, στην απασχόληση που είχαμε κατά διάρκεια της κρίσης έχουν αντισταθμιστεί, τουλάχιστον συνολικά. Ο αριθμός ε, των ανέργων έχει πέσει από 18,6 εκατομμύρια το δεύτερο τρίμηνο του 2014 σε 14,6 εκατομμύρια στο τελευταίο τρίμηνο. Και σε σχέση με το παρελθόν, η αύξηση της απασχόλησης ε, έχει διαπιστωθεί ε, σε διάφορες χώρες και διάφορους τομείς. Σε 16 από τις 19 χώρες ε, της ζώνης του ευρώ είδανε θετική ανάπτυξη της απασχόλησης από τα μέσα του 2014 και η απασχόληση αναπτύσσεται κατά 60 αναπτύσσεται στο 60% των τομέων σε σχέση με 0 στα μέσα του 2014. Αυτά τα, αυτή η βελτίωση της απασχόλησης μαζί με την αύξηση του πλούτου των οικοκυριών ε, στηρίζουν την, ε, τις προβλέψεις ε, για την ιδιωτική κατανάλωση και στις επενδύσεις ε, στις επιχειρήσεις βλέπουμε άνοδο και βλέπουμε και αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων. Τα μέτρα της νομισματικής πολιτικής μας έχουν παίξει ρόλο κλειδί, στηρίζουν και την κατανάλωση και, τις, και τη ζήτηση για επενδύσεις, διασφαλίζοντας ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες. Από τα τέλη του Μαΐου του 2014, τα επιτόκια δανεισμού για ε, μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς έχουν πέσει κατά 120 μονάδες βάσης και για τα νοικοκυριά κατά περίπου 100 μονάδες βάσης. Τα επιτόκια για δανεισμού για τα πολύ μικρά δάνεια που δείχνουν τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, έχουν μειωθεί κατά, κατά σχεδόν 190 μονάδες βάσης και η σημαντική αύξηση στις ε, η σημαντική βελτίωση στι συνθήκε χρηματοδότηση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, διότι αυτέ ε, αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα τη συνολική απασχόληση του ιδιωτικού τομέα στη ζώνη του ευρώ. Αυτή η βελτίωση στι οικονομικέ συνθήκε έχει συνοδευτεί από μείωση της ετερογένειας ε, ανάμεσα στις διάφορες χώρες όσον αφορά τα επιτόκια δανεισμού. Για παράδειγμα, η διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια για τις επιχειρήσεις ε, στις ε, χώρες της ζώνης του Ευρώπου που ε, επλήγησαν περισσότερο από την κρίση σε σχέση με άλλες χώρες έχει στενέψει, η ψαλίδα αυτή έχει ξεν, στενέψει κατά περίπου 100 μονάδες βάσης από τα μέσα του 2014 και παρά την στεναρή οικονομική ανάπτυξη, δεν βλέπουμε ακόμα στον πληθωρισμό να υπάρχει ε, μια ε, τάση προς τα πάνω η οποία να μπορεί να διατηρηθεί. Ε, ο πληθωρισμός ήταν 1,4 τον Οκτώβριο και προβλέπεται να μειωθεί προσωρινά προς το τέλος της χρονιάς, κυρίως λόγω της ενέργειας. Πιέσεις στον πληθωρισμό δεν είναι ακόμα πολύ ισχυρές, διότι και η αγορά ε, εργασίας ε, ακόμη δεν έχει πάρει μπρος και οι βελτιώσει στην αγορά εργασίας που έχουμε παρατηρήσει ε, χρειάζονται χρόνο για να φανούν ως, ανάπτυξη, ως αύξηση των αμοιβών. Και Υπό το φως αυτών των ε, προβλέψεων, ε, κατά την ε, συνάντηση για την νομισματική πολιτική μας τον Οκτώβριο, αποφασίσαμε να αναπροσαρμόσουμε τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής μας. Η αναπροσαρμογή των πολιτικών μας για το διάστημα μετά το τέλος αυτής της χρονιάς στόχο έχει να διατηρήσει την ορμή που έχει σημειωθεί για να διατηρήσουμε πληθωρισμό κάτω από αλλά κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα. Να σας εξηγήσω σύντομα τις τέσσερις βασικές αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο. Καταρχάς, ε, οι βελτιωμένες προβλέψεις και οι μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μας ε, όσον αφορά την ε, σύγκληση των ποσοστών πληθωρισμού μας επέτρεψαν ε, να προσαρμόσουμε και το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων και τον Ιανουάριο του 2018 ανακοινώσαμε ότι οι αγορές περιουσιακών στοιχείων θα συνεχιστούν με ρυθμό 30 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2018 και ενδεχομένως και μετά, ε, όπως και να έχει πάντως, ε, μέχρι το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπιστώσει ότι υπάρχει μόνιμη ε, προσαρμογή όσον αφορά τον πληθωρισμό. Δεύτερον, όσον αφορά την πολιτική επανεπενδύσεων, δηλώσαμε ότι το σύστημα του ευρώ θα επαναεπενδύει τις πρωτογενείς πληρωμές από αξιόγραφα που λήγουν για για ένα ε, εκτενές χρονικό διάστημα μετά το τέλος των ε, αγορών περιουσιακών στοιχείων και αυτό θα συμβάλλει και ε, σε καλές συνθήκες όσον αφορά τη ρευστότητα και σε μια κατάλληλη νομισματική πολιτική. Και θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι παρήχαμε και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα ποσά ε, αγοράς για κάθε στοιχείο του συστήματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Οι πολιτικοί μας να συνεχίσουμε να επενεπενδύουμε τα κέρδη από αυτά τα αξιόγραφα έχουν γίνει πιο σημαντικά διότι αυξάνεται και το μέγεθος του χαρτοφυλακίου μας. Και η ιστοσελίδα μας αναφέρει όλα τα αποτελέσματα ε, σχετικά με τα ποσά που αναμένονται για το επόμενο δεκάμινο. Τρίτον, ε, όσον αφορά τα επιτόκια, τα διατηρήσαμε όσοι είχαν και επαναλάβαμε ότι περιμένουμε ε, τα ε, βασικά μας επιτόκια να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα για πολύ χρονικό διάστημα και αφού έχουμε ε, περάσει τον ορίζοντα του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Αυτά αποτελούν βασικά στοιχεία της νομισματικής μας πολιτικής αυτή τη στιγμή. Και όταν λέμε ότι θα διατηρηθούν για πολύ διάστημα μετά την ελήξη του σχετικού προγράμματος, αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν σημαντικό παράγοντα ενδυνάμωσης ώστε οι αγορές περιουσιακών στοιχείων να ε, μπορέσουν να έχουν τον πλήρη τους αντίκτυπο. Τέλος, ε, αποφασίσαμε ότι οι ε, εργασίες αναχρηματοδότησης μας θα συνεχιστούν για όσο είναι απαραίτητα και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2019. Και αυτό θα διασφαλίσει ομαλή εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής μας ενώ θα διασφαλίζει και ευνοϊκές συνθήκες στις ε, αγορές κεφαλαίων στην ζώνη του ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπέρανε στο τέλος της τελευταίας συνάντησης ότι η στήριξη νομισματικής πολιτικής που παρέχουμε σήμερα προέρχεται από το συνδυασμένο αποτέλεσμα των επιπλέον αγορών περιουσιακών στοιχείων, ε, το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων που έχουν ε, συγκεντρωθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό στο παρελθόν ε, και οι επανεπενδύσεις ε, των αγράφων που λήγουν, καθώς ε, και οι κατευθυντήριε γραμμές που δίνουμε για τα επιτόκια. Τα μέτρα αυτά θα διατηρήσουν τις παρούσες συνθήκες χρηματοδότησης και θα διασφαλίσουν επαρκή βαθμό κινήτρων που είναι απαραίτητα ώστε να έχουμε πληθωρισμό κοντά σε αλλά κάτω από το 2%. Να αναφερθώ τώρα στα ισοζύγια target. Το target 2 είναι το σύστημα ε, διακανονισμού σε πραγματικό χρόνο του ζώνης του ευρωμέσου, του οποίου πληρωμές σε ευρώ μπορούν να διεκπεραιώνονται ε, με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ τραπεζών ε, και εντός μιας χώρας και διασυνοριακά. Παρέχει υποδομή που χρησιμοποιείται για τον διακανονισμό για διεκπαιρέωση πληρωμών ε, σε μια ευρία γκάμα ε, συναλλαγών ε, που έχουν να κάνουν με τις χρηματοπιστωτικές αγορές, συναλλαγές μεταξύ τραπεζών και πληρωμές πελατών. Πέρσι το Target 2 επεξεργαζόταν κατά μέσο όρο 342.000 πληρωμές την ημέρα και αντιπροσώπευε έτσι καθημερινά αξία 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό παίζει ρόλο κλειδί στην διασφάλιση της ε, ομαλής ε, νομισματικής πολιτικής, ε, την σωστή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Με στήριξη της δημοσιονομικής ολοκλήρωσης και την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής μας, το Target 2 αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της νομισματικής μας ένωσης στο σύστημα αυτό κάθε τράπεζα έχει έναν πιστωτή και έναν οφηλέτη σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, που εξετάζει ε, τα χρήματα που μπαίνουν και βγαίνουν ε, από κάθε χώρα για λογιστικούς λόγους. Τα ισοζύγια target λοιπόν απλά αντικατοπτρίζουν τον διακανονισμό διασυνοριακών πληρωμών που γίνονται μέσω του target 2. Οι πληρωμές που γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων επίσης ε, γίνονται μέσω του Target 2. Και η εφαρμογή του συστήματος ε, αγοράς περιουσιακών ε, στοιχείων διαχωρίζεται από τις λειτουργίες αναχρηματοδότησης ε, που γίνονται. Μάλιστα το 80% των ε, συνολικών ε, αγορών έχουν γίνει από παράγοντες των χρηματοπιστωτικών αγορών που δεν βρίσκονται στην ίδια χώρα με την κεντρική τράπεζα που αγοράζεται περιουσιακά στοιχεία και έτσι επηρεάζονται τα ισοζύγια target. Επιπλέον, οι πολιτές των περιουσιακών στοιχείων που αγοράζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό μπορούν να επανεπενδύσουν τα κέρδη και έτσι να έχουμε ε, επανεξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου τους. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αλλαγές ε, στα ισοζύγια target, ακολουθώντας τη λογική που μόλις σας περιέγραψα. Παρόλα αυτά, το Target 2 ε, είδαμε ότι έχει συμβάλει στην ομαλή εφαρμογή των ε, μέτρων νομισματικής ε, πολιτικής μας ε, και, στην, και στο να υπάρχουν ομαλές συνθήκες χρηματοδότησης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μας. Να κλείσω λέγοντας ότι ε, στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα είναι να διατηρηθεί η σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Και αυτή είναι η καλύτερη συμβολή που μπορούμε να κάνουμε ε, για την ευημερία των συμπολιτών μας. Να διασφαλίσουμε δηλαδή τη σταθερότητα ε, των τιμών, διότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση ώστε να έχουμε ισορροπημένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη. Αλλά αυτό δεν αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση. Το να έχουμε Εξισορροπημένη ανάπτυξη σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει η ζώνη του ευρώ να γίνει πιο ανθεκτική στους κινδύνους όποτε αυτοί εμφανιστούν. Και οι παρούσες οικονομικές προβλέψεις μας παρέχουν μία μοναδική ευκαιρία να μειώσουμε την πιθανότητα κλειδονισμών ενισχύοντας τις οικονομικές δομές των κρατών μελών με δράσεις πολιτικής και σε δημοσιονομικό και σε διευθυντικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, Αυξάνοντας την αθεκτικότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωση, θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε το θεσμικό μας πλαίσιο, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε και να διαχειριστούμε ε, κλειδονισμού στο μέλλον. Και γι' αυτό επικροτώ τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις συζητήσεις αυτές ε, και τις ε, ανανεωμένες προσπάθειες ε, των ε, ηγετών της ζώνης του ευρώ να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, όπως για παράδειγμα αυτό αντικατοπτρίζεται στην πρόσφατη συνάντηση του Eurogroup. Και στο πνεύμα αυτό προσβλέπω στην διάσκεψη κορυφής για το ευρώ που θα έχει ως αντικείμενο την διακυβέρνηση της, ζώνης, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας. ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Ντράγκη. Θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Κυρία Ντελάγκε έχει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρο, ευχαριστώ τον Πρόεδρο Ντράγκη για την παρουσία του εδώ που είναι διατεθειμένος να δώσει απαντήσεις σε θέματα σημαντικά για την Οικονομική Επιτροπή. Τα κόκκινα δάνεια τώρα. Εσείς ε, έχετε ε, περιγράψει σαν ένα σημαντικό βάρος αυτό το φαινόμενο για το τραπεζικό σύστημα. Ξέρω επίσης ότι έχετε προτείνει αρκετά μέτρα σαν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα έχετε και σύντομα μία συνάντηση για το θέμα αυτό. Το ίντις λοιπόν και το θέμα της μείωσης των κινδύνων γενικά συνδέονται μεταξύ τους όχι μόνο σε επίπεδο περιεχομένου και ουσίας αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Πώς μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε με το ίντις γιατί αυτό ακριβώς θέλουμε αν ε, υπάρχει πολύ μεγάλος δισταγμός ε, σε πολλές χώρες σχετικά με τα NPL, στα κόκκινα δάνεια. Ε, και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί ε, ο σωρός εισαγωγικά των MPL ε, γιατί προς το παρόν περιμένει σαν να περιμένουμε ότι από ένα θαύμα θα εξαφανιστεί από μόνο του το πρόβλημα αυτό. Και σε ποιο βαθμό το θέμα αυτό τίθεται και σε διεθνές επίπεδο και επηρεάζει το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς σαν εισηγητές και συνεισηγητές στα πλαίσια του ίντις. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις παρεμβάσεις σας μέχρι τώρα και για τις απαντήσεις σας από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπατε, τα NPL και το ίντις συνδέονται μεταξύ τους, είναι αλληλέμβετα. Είπαμε για το ίντις να πω ότι στην ουσία εμείς καλωσορίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγοντας όμως ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ποιος είναι ο τελικός στόχος, η πλήρης κάλυψη αν θέλετε. Μπορεί να έχουμε έναν στόχο τελικό, αλλά στον στόχο θα φτάσουμε με σταδιακό τρόπο. Κάθε βήμα προόδου όμως θα πρέπει να είναι σαφέστατα ποσοστοκοποιημένο και ε, κατανοητό με, ξεκάθαρα, ε, με ξεκάθαρες διαστάσεις και σταθμά. Δεν θα πρέπει να είναι μια απλή αναβολή αν θέλετε της επιδίωξης μιας κάποιας λύσης το ίδις παραμένει ένας βασικός πυλώνας του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη. Πάντως η μείωση των κινδύνων και η διανομή αν θέλετε των κινδύνων παραμένει ένα από τα χαρακτηριστικά της πρακτικής ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το πρόβλημα αυτό των κόκκινων δανείων είναι ένα πρόβλημα το οποίο εξακολουθεί ε, να παραμένει. Τα ακούσατε και από την κυρία Νουή. Είναι κυρίως θέμα εποπτείας. Απαιτεί μια κοινή προσπάθεια, το έχω πει και εγώ, και από τις διαχειριστικές ομάδες των τραπεζών και από τις εποπτικές αρχές και από τις κυβερνήσεις και από τους νομοθέτες έτσι ώστε να διασφαλιστεί ένα συνολικό νομικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει στα NPL να γίνουν εμπορεύσιμα και να εξαφανιστούν σε κάποια φάση αν θέλετε. Λοιπόν, τώρα βέβαια τα βήματα τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα ε, ασχολούνται με τα καινούργια NPLs και όχι με την κληρονομιά των κόκκινων δανείων ε, που οδήγησε σε καταστάσεις που χαρακτήρισαν ε, τα τελευταία χρόνια πριν φτάσουμε στην περίοδο της οικονομικής ανάπτυξης. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα θέματα τα κληρονομικά σε εισαγωγικά πριν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των κόκκινων δανείων από εδώ και πέρα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Γκουαλτιέρη. Και εγώ και άλλοι ενθυμούμεθα τα σοφά λόγια που μας είχατε πει για την κοινότητα των προσπαθειών από όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και τις κυβερνήσεις και να πω ότι ο διάλογος με την κυρία Νουή και τα συμπεράσματα ήταν πάρα πολύ χρήσιμος. Είναι σαφές ότι απαιτείται να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα όταν αυτό θεωρούνται απαραίτη, θεωρείται απαραίτητο. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων βέβαια του κάθε οργάνου και του κάθε επίπεδου και εδώ ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καθοριστικός ε, γιατί θα βοηθήσει καταρχάς να ποσοστικοποιήσουμε ακριβώς τις δυνατότητες που έχει κάθε συμβαλόμενο μέρος. Η κυρία Μπερές για την ομάδα των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα επανέλθω σε αυτή τη συζήτηση ε, για το EMPL και το EDIS, ε, παρά το ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε τη συζήτηση και να αναρωτιόμαστε για σε ποιες συνθήκες ε, η εφαρμογή αυτών των δύο πυλώνων της Τραπεζικής Ένωσης, είτε από την πλευρά της επίβλεψης είτε από την πλευρά της εξυγίανσης, δεν κατάφερε να μας οδηγήσει σε ποσοτικοποιημένη πρόοδο τεράστια όσον αφορά τη μείωση κινδύνου. Το ερώτημά μου, θα σας το πω, κατόπιν ενός, ζητήματο, ζητήματος που μας είχατε αναφέρει στην περασμένη ανταλλαγή απόψεων ε, κατά το δημοκρατικό μας διάλογο μαζί σας. Ο συνάδελφος Πολ Τόγκ μας είχε, σας είχε κάνει μια ερώτηση σε σχέση με τους μισθούς. Θυμάστε ότι μιλήσατε για την αύξηση, το ρυθμό αύξησης των μισθών στις χώρες ε, στις οποίες ε, η, ε, φαίνεται να έχει γίνει μια αλλαγή στην οικονομική ανάκαμψη ε, της και τις οικονομικές πολιτικές τους, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να, διευκολύνει ε, τη νομισματική πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι είναι μία συζήτηση που θα απασχολούσε βέβαια με τον οικονομολόγο, αλλά και όσοι ασχολούνται με τα τραπεζικά ε, μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή. Όπως επίσης υπάρχει και το θέμα της μείωσης της, ε, ε, της συνδικαλιστικής ικανότητας των εργαζομένων. Πώς θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια αύξηση των μισθών. Είναι μια συζήτηση που κάναμε και με τον Κάλλος Κώστα, τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Πορτογαλίας. Με διαφορετικό σενάριο βέβαια. Η ιδέα είναι ότι η παγκοσμιοποίηση άλλαξε τις συνθήκες καθορισμού των μισθών και συνεπώς αντί Αντί να ευημερούμε λοιπόν σύμφωνα με τους παλιούς κανόνες, ίσως θα μπορούσαμε να δούμε ε, ποιες, ποια, είναι, ποια είναι τα θεμέλια της νομισματικής πολιτικής. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν συζητάτε καθόλου στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόσφατη πολιτική μας, ε, η τα πρόσφατα μέτρα νομισματική, νομισματικής πολιτικής μας αντικατοπτρίζουν ε, πολλές αξιολογήσεις ε, του Διοικητικού Συμβουλίου, την πεποίθηση ότι ο πληθωρισμός θα μετακινηθεί και θα φτάσουμε όντως κάποια στιγμή στο στόχο μας λόγω της ανάκαμψης και λόγω της αύξησης της απασχόλησης. Όμως, όταν περνάμε ε, στην πλευρά του πληθωρισμού και τη σχετική αξιολόγηση, βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός είναι πολύ περιορισμένος και ο λόγος που είναι περιορισμός είναι το γεγονός ότι υπάρχει ο ο ε, πληθωρισμός που έχει να κάνει με τις αλλαγές των τιμών ε, της ενέργειας και αυτό παραμένει περιορισμένο και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός σε μη ονομαστική αύξηση των μισθών. Αυτό συμβαίνει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε σύγκριση τώρα με άλλους ε, επιχειρηματικού κύκλους στο παρελθόν, η σχέση των ονομαστικών μισθών ε, με την κάλυψη των κενών, την αύξηση και τη βελτίωση των, της αγοράς εργασίας, ε, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, 4 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης σε 4 χρόνια. Δεν είναι λίγο αν το σκεφτείτε όλες, ε, όλη αυτή η αξιοσημείωτη αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας έγινε σε... Ε, σε σχέση, ε, σε συνδυασμό με ποσοστά συμμετοχής αυξημένα. Ε, υπήρχε επίσης και το θέμα της κρίσης λόγω της ε, προσέλευσης των μεταναστών, όπως επίσης και τη συμμετοχή των γυναικών. Πρόκειται για επίπεδα που είναι άνευ προηγουμένου η συμμετοχή των μεγαλύτερης ηλικίας επίσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ ψηλό ποσοστό ε, με αυτούς λοιπόν τους ε, νέους παίκτες στην αγορά εργασίας παρόλα αυτά υπήρχε μια σημαντική μείωση στην ανεργία και όλα αυτά ε, δείχνουν ότι είναι μια πολύ επιτυχημένη εμπειρία. Δεν θεωρούμε ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη ονομαστική αύξηση των μισθών θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι η παγκοσμιοποίηση ο λόγος ε, ή ότι ε, δεν προέρχεται τόσο, δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της Ευρωζώνης αλλά είναι ένα παγκόσμιο ε, φαινόμενο. Δεν θεωρούμε όμως ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος λόγος. Το κενό output στον υπόλοιπο κόσμο είναι συνδεδεμένο και με το δικό μας, οπότε λογικά θα θεωρούσαμε ότι θα μπορούσε να ε, συνδέεται. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ένα, μια περίοδος ε, χαμηλού ε, πληθωρισμού. Φυσικά κάποιες, θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες υπαναχωρήσεις και θα μπορούσαμε έτσι να ε, ληφθεί υπόψη στι επόμενε διαπραγματεύσεις αυτή η προβληματική του χαμηλότερου πληθωρισμού μετά από μια μεγάλη περίοδο ανεργίας και μεγάλες ε, δύσκολες συνθήκες στην αγορά εργασίας ε, η στρατηγική ως προς την απασχόληση είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια στην απασχόληση και όχι τόσο αύξηση των μισθών. Και αυτό είναι ένας άλλος λόγος ε, να μην ξεχνούμε ότι η παραγωγικότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και αυτό είναι ένας τρίτος διαρθρωτικός λόγος. Σε γενικές γραμμές όμως, όσον αφορά τους δύο πρώτους λόγους κυρίως, ε, θεωρούμε ότι είναι κάτι σοβαρό, αλλά είναι κάτι το περαστικό. Ε, επειδή υπάρχει υποστήριξη από την νομισματική μας πολιτική, από την νομισματική μας πολιτική και υπάρχει συνέχεια, γιατί είπα και, ε, είπα και προηγουμένως ότι υπάρχει μία αύξηση η οποία φαίνεται να μην ε, ε, διακόπτεται, να είναι αδιάκοπη, θεωρούμε ότι θα συνεχίσει προς αυτή την ε, κατεύθυνση. Όλες αυτοί, όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες ε, που αφορούν για παράδειγμα τις διαπραγματεύσεις για τους μισθούν και η προτίμηση υπέρ της ασφάλειας στην απασχόληση που είπα ότι την έχουμε, θεωρούμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των μισθών. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, αξιολογώντας το γεγονός ότι ε, υπάρχει χαμηλός πληθωρισμός ε, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο και πιστεύουμε ότι ως προς το πληθωρισμό κινούμεθα όντως προς το στόχο μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τράκη. Ε, θα μιλήσω γερμανικά. Μία σύντομη παρατήρηση καταρχάς. Μ' ακούτε? Μία σύντομη παρατήρηση σχετικά με την απάντησή σα. Είπατε ότι 4 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πώς το ξέρουμε ότι τις ε, δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν έχουν δημιουργηθεί και θέσεις απασχόλησης ε, εκτός ε, της ζώνη εργασίας και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι εντό τη Ευρωζώνης θα μπορούσατε, ε, νομίζω θα, θα έπρεπε να έχουμε πιο εμπεριστατωμένες πληροφορίες, αλλά δεν θα ήθελα να απαντήσετε σε αυτό, αλλά στο εξή. Στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επενδύσει 1,6 εκατομμύρια σε ομόλογα χωρών ε, της ζώνης του ευρώ. Η ερώτησή μου είναι πολύ απλή. αληθεύει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, είναι πάροχος πιστώσεων για χώρες της ζώνης του ευρώ και μάλιστα πολύ σημαντικός ε, τέτοιος πάροχος πιστώσεων. Uh, Ζητώ συγγνώμη, δεν κατάλαβα τη δεύτερη ερώτησή σας. Ο κύριος Λούκε, η ερώτησή μου είναι, έχω δίκιο εάν πω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μεγάλος και μόνιμος πιστωτής των κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ. Η απάντηση στη δεύτερη ερώτησή σας είναι όχι. Διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνολικά έχει αγοράσει, δεν θυμάμαι τώρα το ποσοστό, αλλά 10, 15 με 20% των ε, συνολικών αξιογράφων. Ε, δεύτερον, ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα έχει αγοράσει αυτά σε ε, παράγωγε αγορέ, δηλαδή από άλλου, όχι από τι κυβερνήσει που τα εξέτωσαν. Και όσον αφορά την πρώτη σα ερώτηση. Έχω μια δεύτερη ερώτηση. Δεν χρειάζομαι απάντηση στην πρώτη μου ερώτηση. Όπως ήδη είπα. <laughs> Μία τρίτη ερώτηση θα ήθελα να θέσω αν μου επιτρέπετε και πάλι στα γερμανικά αν μου επιτρέπετε. Η διαφορά ανάμεσα στις ε, πρωτογενείς και δευτερεύουσες αγορές, ε, παράγωγες αγορές, είναι γνωστή σε μένα. Αλλά Τη στιγμή που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτά τα ομόλογα, δεν παίζει ρόλο που τα αγόρασε, εφόσον τα έχει, δίνει πιστώσει σε χώρε τη ζώνη του ευρώ. Και η ερώτησή μου είναι, αναφερθήκατε εσεί στο μέγεθο των στον όγκο των αξιογράφων. Για κάποια κράτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αγοράσει το 350% των αξιογράφων που εξέδωσαν ε, ως νέα ομόλογα τα κράτη στο διάστημα 2015-2017. Ε, το 52%, συγγνώμη, το 52%. Και αυτό όπως συνάδει με την απαγόρευση της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού των κρατών μελών. Είναι πολύ απλό αυτό. Ε, δεν παραβιάζουμε τον κανόνα αυτό. Ε, απλά συμμορφούμαστε με την εντολή μας σύμφωνα με την ε, Ευρωπαϊκή Συνθήκη και με τον νόμο. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση στη δεύτερη ερώτηση. Θέλετε να απαντήσω τώρα στην πρώτη σας ερώτηση. Η πρώτη σας ερώτηση είναι πώς γνωρίζουμε. Ε, πώς να μην το γνωρίζουμε. Το ξέρουμε διότι Χάρη στις οικονομικές συνθήκες που έχει δημιουργήσει η οικονομική πολιτική ήταν δυνατή η ανάπτυξη. Αυτή ήταν η βασική πολιτική εδώ και πολλά χρόνια. Ενώ πριν δεν υπήρχαν καθόλου πολιτικές. Μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, αλλά έχουμε πολλά ενδεικτικά στοιχεία. Ότι η πολιτική έχει οδηγήσει στην ανάκαμψη που βλέπουμε σήμερα. Δέκα δευτερόλεπτα. Κύριε Ντράγκη, στα αγγλικά θα μιλήσω. Σας ρώτησα εάν παραβιάσατε την εντολή σας ή εάν μπορείτε να εξηγήσετε ότι δεν πρόκειται για συμμόρφωση ε, των, ε, για παραβίαση της συμμόρφωσης της εντολής σας εφόσον αγοράσετε το 250% λέει ε, των αξιογράφων. Όχι, όχι, δεν την παραβιάσαμε. Συμμορφωθήκαμε με την εντολή μας. Ε, μείναμε εντός των ορίων που ε, θέσαμε ήδη από την αρχή του προγράμματος. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Νομίζω ότι και ο κύριο Λούκη γνωρίζει πολύ καλά τη διαφορά ανάμεσα στο Ευρωσύστημα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τρεμόσα, παρακαλώ. Καλώς ήρθατε, Πρόεδρε Ντράγκη, στην Επιτροπή μας. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη. Τον Ιανουάριο του 2018 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αρχίσει να μειώνει το EQ, το QE συγγνώμη, έτσι ώστε σιγά σιγά Κάτι όμως το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στις πιο, θα έλεγα, χρεωμένες χώρες. Τι θα προτείνατε για τις χώρες αυτές όπου το έλλειμμα τους είναι άνω του 3% του ΑΕΠ. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μια νέα ύφεση. Τώρα για το ίντις συζητάμε το θέμα της εγγύησης των καταθέσεων, πάντα το έχετε υποστηρίξει. Θα ήθελα να μας πείτε κύριε Ντράγκη πώς βλέπετε εσείς πώς θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Τι είναι σημαντικό έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Πώς μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους ε, επενδυτές ότι το ίντις θα δουλέψει καλά γιατί έχουν υπάρξει κάποια προβλήματα στο παρελθόν σε σχέση με Ιταλικές τράπεζες και με την Ισπανική Banco Popular. Να ξεκινήσω με τη δεύτερη ερώτησή σας, λέει ο πρόεδρος Ντράγκη. Η παρατεταμένη συζήτηση την οποία είχαμε για το Ίντις έπεισε τους πάντες ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόματα και άμεσα γιατί πρέπει να επαληθευθούν ορισμένες συνθήκες, προϋποθέσεις και από τη μία η μείωση του κινδύνου και από την άλλη η κατανομή των κινδύνων πρέπει να πηγαίνουν με εναρμονισμένο τρόπο. Πρέπει να υπάρξουν δηλαδή κάποια εναμονισμένα χαρακτηριστικά κρίσιμα για, την, για το ευρωπαϊκό πιστοτικό σύστημα. Αν έχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας οι διάφορες χώρες, αυτό σημαίνει ότι η Ένωση η Τραπεζική δεν είναι ολοκληρωμένη και η άλλη εναρμόνιση η οποία είναι απαραίτητη είναι η διαδικασία για την εξυγίανση. Η καθεστώτα εξυγίανσης είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και η πιστοτική ένωση. Πάντως το θέμα της μείωσης των κινδύνων έχει να κάνει και με τα NPL, τα κόκκινα δάνεια τα οποία συζητήσαμε ήδη και εν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρατηρεί ότι όλα αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούν να επιτευχθούν σταδιακά χωρίς να χάσουμε τον τελικό στόχο από μπροστά μας, ε, μια πλήρη κάλυψη των καταθέσεων και να είμαστε βέβαιοι ότι οδεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή και η πορεία προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται πάντα, να είναι σαφής και προσμετρήσιμη σε κάθε στιγμή και φάση. Τώρα οι χώρες είναι έτοιμες, είναι σε θέση για την πολιτική μας μείωση των κινήτρων, να το πω έτσι. Καταρχάς δεν το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Η αναστάθμιση την οποία στην ουσία εμείς αποφασίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα όταν την ανακοινώσαμε, αυτό επηρέασε τις χρηματαγορές κατά μηδενικό τρόπο. Ήταν ακριβώς κάτι το οποίο είχε μετρηθεί σε σχέση με την βελτίωση και τη στάθμιση των ρυθμών βελτίωσης της οικονομίας. Και παρόλα αυτά οι, οι μηνιαίες ροές μειώθηκαν στα 30 από τα 60 που ήταν. Συνεπώς λοιπόν υπήρξε μια ουσιαστική μείωση χωρίς προβλήματα. Η μείωση λοιπόν των κινήτρων η οποία θα συνεχιστεί εφόσον και οι συνθήκες το επιτρέπουν τότε θα γίνει στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος το οποίο θα μας επιτρέψει να μην αναμένουμε περαιτέρω αλλαγές. Να πούμε ότι η εντολή μας είναι η σταθερότητα των τιμών και όχι η δημοσιονομική στήριξη προς τις κυβερνήσεις. Και τέλος, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο σταθήκατε και με το οποίο θα συμφωνήσω πλήρως. Να πω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή πλέον, όχι μόνο να να περάσουμε στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, τις δομικές που απαιτούνται, αλλά να βελτιώσουμε επίσης και τις φάσεις ε, σε επίπεδο δημοσιονομικό. Και ακριβώς ε, το, ο λόγος για τον οποίο θα συμβεί αυτό είναι ότι οι ε, χώρες θα πρέπει να αποκτήσουν ένα κάποιο χώρο αν θέλετε πολιτικής ε, παρέμβασης σε περίπτωση που υπάρξει μια κάποια ύφεση στο μέλλον ή μια κρίση στο μέλλον. Ο κύριος Παπαδημούλης. Ε, κύριε Ντράγκη, θα σας μιλήσω στα ελληνικά. Εδώ ε, σας καλωσορίζω και πάλι στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ορισμένα πράγματα. Το πρώτο αφορά στη χώρα μου την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετέχει στους θεσμούς που εκπροσωπούν τους δανειστές. Και τώρα τελευταία ακούμε θετικές προβλέψεις από την Κομισιόν, από τον ESM για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, για την πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Θα ήθελα να μου δώσετε τις δικές σας εκτιμήσεις της ECB για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, για την προοπτική ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και ιδιαίτερα τη γνώμη σας για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τις αποκαλύψεις αυτής της σκανδαλώδους μεγάλης φοροδιαφυγής μέσω των Paradise Papers. Ο Επίτροπος Μοσκοβισή πριν μία εβδομάδα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου μίλησε για βαμπύρ της φοροδιαφυγής και είπε πως πρέπει να ληφθούν μέτρα διαφάνειας, ανταλλαγής πληροφοριών, φορολογικής εναρμόνισης, διότι εκτός από τους φορολογουμένους πλήττεται και η ευρωπαϊκή οικονομία μέσω αυτής της σκανδαλώδους αποφυγής πληρωμής φόρων από τους υπερπλουσίους. Θα ήθελα την εκτίμηση τη δική σας, την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέναντι σε αυτήν τη φοροδιαφυγή και στο πώς μπορεί αυτή να αντιμετωπιστεί. Και η τελευταία μου ερώτηση αφορά την έκθεση που δόθηκε πριν λίγες μέρες στη δημοσιότητα από ένα θεσμικό όργανο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο αξιολόγησε την πορεία εφαρμογής των μνημονίων στη χώρα μου την Ελλάδα, εντόπισε πολλά λάθη στο σχεδιασμό με αρνητικές κοινωνικές συνέπειες και ένα έλλειμμα αξιολόγηση των κοινωνικών συνεπειών. Στην έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνει ότι δεν μπορεί να αξιολογήσει το ρόλο που έπαιξε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα ελληνικά προγράμματα γιατί αρνηθήκατε να δώσετε τις πληροφορίες που σας ζήτησε. Μπορείτε να μου σχολιάσετε αυτή την ε, επισήμαση. Πώς απαντάτε στην κριτική του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρώπης. Thank you. Ευχαριστώ. Για το πρώτο ερώτημα που αφορά την βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και πράγματι έχει βελτιωθεί συνολικά η κατάσταση σε μεγάλο βαθμό και από απόψε ως απασχόληση και από απόψε ως ΑΕΠ η συνεχής εφαρμογή πολλών μέτρων που παρουσιάστηκαν κατά την τρίτη αξιολόγηση ήδη καρποφορεί. Βλέπουμε επίσης ε, ότι οι αλλαγές ε, φαίνονται και ε, στο χρέος το ελληνικό που είδαμε μείωση των spreads επίσης βλέπουμε και μια θετική ανταπόκριση των αγορών στο, στα μέτρα debt swap ήδη έχει βελτιωθεί η ρευστότητα του δημοσίου χρέους, κάτι το οποίο φαίνεται, φαίνεται στην ανταπόκριση των αγορών. Θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία αναλογία 17,1% που είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό ποσοστό Πρέπει βέβαια οι τράπεζες να σταθεροποιήσουν την κατάστασή τους, ε, γιατί αυτή τη στιγμή η κατάσταση των καταθέσεων ε, έχει μεν σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει επανέλθει στα πρώτης κρίσεως επίπεδα. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, Η φορολογία, όπως γνωρίζετε, δεν είναι κάτι που παρακολουθείτε και δεν αποτελεί τμήμα του δικών μας καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την φόρο διαφυγή και την φόρο αποφυγή. Ε, βεβαίως συμφωνούμε με ό,τι θα προτείνουν οι συνομοθέτες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς αυτό. Εμείς πάντοτε υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις προτάσεις των συνομοθετών ε, ως προς αυτό. Για το τελευταίο σας ερώτημα τώρα, αναφερθήκατε στο ελεγκτικό συνέδριο και την έκθεσή του. Καταρχάς, έχω ένα γενικό σχόλιο να κάνω. Το η εντολή του ελεγκτικού συνεδρίου περιορίζεται στην ανάλυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της διαχείρισης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όταν λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο κάνουν ερωτήσεις που υπερβαίνουν αυτήν την εντολή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να απαντήσει, ειδικότερα όταν οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με τα στοιχεία που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, στο Eurogroup, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συνεπώς δεν υπάρχουν αποδυτικά στοιχεία στο πλαίσιο της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου που θα υποστήριζαν αυτόν τον ισχυρισμό που κάνατε προηγουμένως ότι υπήρξαν σφάλματα και ούτω καθεξής. Η αξιολόγηση κεφαλαιακών απαιτήσεων πάντοτε βασίζεται στις μακροεποθέσεις που είναι διαθέσιμες ε, όταν γίνονται τεστ ε, αντοχής επίσης ε, εννοώ δηλαδή ότι εντάξει προφανώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να συνεργαστεί και να συνεχίσει να έχει μια συνεργασία καλή με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Νομίζω ότι είπα ό,τι είχα να πω εν προκειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φίλιπ Λάμπερτς. Καταρχάς, ως προς τη δυναμική των μισθών. Όταν βλέπω το ποσοστό απασχόλησης όσον αφορά ε, την χρήση, την ικανότητα είναι 63% στο Βέλγιο, είναι 53% στη χώρα σας στην Ιταλία. Με τόσο ε, τεράστια υποαπασχόληση, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση που δεν αυξάνονται οι μισθοί. Είναι προφανές. Μάλιστα, ε, η Πάτε ότι θα χρειάζεται, ο κόσμος χρειάζεται σταθερότητα της απασχόλησης. Προφανώς, όλος ο κόσμος προτιμά μια σταθερότητα στην απασχόληση. Μιλήσατε για την αύξηση του πλούτου των οικοκυριών. Τι μπορείτε να μας πείτε για, τον, για την κατανομή αυτής της αύξησης. Εποφελείται όλος ο κόσμος ή ε, βλέπουν κάποιοι το πλούτο τους να μειώνεται και ο ε, πλούτος κάποιων άλλων αυξάνεται και έχει να, μπορούμε να το συγκρίνουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, στις οποίες τα τελευταία 10 χρόνια το 99% της αύξησης του πλούτου πηγαίνει στο 1% του πληθυσμού. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Εσείς ε, έχετε μία ε, πολύ καλή θεώρηση του ευρύτερου ε, χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τι αδυναμίες θεωρείτε ότι υπάρχουν στο σύστημα, στο σύστημα εντός της Ευρωζώνης αλλά και εκτός της Ευρωζώνης που θεωρείτε ότι επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό ε, την κατάσταση των χωρών της Ευρωζώνης. Τι είναι αυτό δηλαδή που σας κρατά ξύπιο τη νύχτα όσον αφορά τη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερικοί παράγοντες. Ευχαριστώ. Uh, Όσον αφορά την πρώτη σας παρατήρηση, συμφωνώ απολύτως. Μάλιστα στην απάντησή μου σχετικά με το γιατί οι ονομαστικοί μισθοί δεν μειώνουν το κενό παραγωγής είναι και αυτός ένας λόγος. Εάν μετρήσουμε την ανεργία με βάση το U6, αυτό που είπατε εσείς, την ποιότητα δηλαδή των θέσεων απασχόλησης, βρίσκουμε και άλλη μια εξήγηση για το γιατί οι ονομαστικοί μισθοί δεν ε, έχουν προσαρμοστεί ανάλογα. Ταυτόχρονα, όσο παρέχεται ε, νομισματική ε, στήριξη και αυτό θα φαίνεται τους ε, μισθούς. Ε, θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα αυξηθούν και οι ονομαστικοί μισθοί. Ε, θα μπορούσε να δώσει κανείς μια απλουστική, μια απλοϊκή απάντηση λέγοντας ότι φταίει η παγκοσμιοποίηση ή η ψηφιοποίηση. Αλλά δεν είναι αυτή η βασική λόγη. Η βασική λόγη είναι αυτή που αναφέρατε εσείς και αυτή που ανέφερα εγώ πριν. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να αναπροσαρμόζουμε την νομισματική πολιτική ώστε να δούμε αυτήν την βαθμία βελτίωση στην αγορά εργασίας μέχρι το βαθμό που θα δούμε αλλαγή στους ονομαστικούς μισθούς. Όσον αφορά την κατανομή του πλούτου, δεν το είπατε και είμαι βέβαιος ότι δεν το λέγατε, αλλά να καταστήσω σαφές ε, σχετικά με την ε, ανισότητα, αυτό δεν είναι αλήθεια. Φυσικά, αν αγοράζει κανείς ε, περιουσιακά στοιχεία, οι τιμές ε, ανεβαίνουν. Ε, οι κάτοχοι των περιουσιακών στοιχείων ε, γενικά είναι πλούσιοι άνθρωποι. Ε, έτσι μπορεί να φαίνεται σαν να επιδεινώνεται η κατανομή του πλούτου, αλλά μπορεί να βελτιώνεται η αγορά εργασία, για παράδειγμα. Και εδώ ακριβώ έχουμε τη βασική πηγή και τον πιο βασικό λόγο για την ανισότητα στον πλούτο και στα εισοδήματα, την ανεργία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ουσιαστικά βελτίωση ε, όσον αφορά την κατανομή του πλούτου και την ανισότητα εισοδημάτων. Μάλιστα, βραχυπρόθεσμα μπορεί να φαίνεται ότι πετυχαίνουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, ότι έχουμε περισσότερη ανισότητα, αλλά μακροπρόθεσμα βλέπουμε ότι αντισταθμίζονται αυτά τα ε, βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. επιπλέον οι επιπτώσεις ε, της ε, νομισματικής πολιτικής μας ε, στις τιμές των κατοικιών έχει βελτιωθεί. Βλέπουμε ότι μειώνεται η ανισότητα όσον αφορά τον πλούτο, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους που μπορούν πιο εύκολα έτσι να αγοράσουν μια κατοικία. Είναι η κατάσταση τόσο κακή όσο είναι και στι ΗΠΑ. Η απάντηση είναι όχι. Η κατανομή πλούτου και εισοδημάτων στην Ευρώπη, τουλάχιστον στην υπηρετική Ευρώπη, είναι καλύτερη. Έχουμε βέβαια διαφορετικό ε, κοινωνικό μοντέλο το οποίο ε, έχει προστατεύσει την κατάσταση, παρότι είδαμε ότι η δραματική αύξηση της ανεργίας κατά διάρκεια της κρίσης ε, έχει επιδεινώσει ε, την κατάσταση. Και όσον αφορά την ε, δημοσιονομική σταθερότητα. Παρακολουθούμε στενά τα επιτόκια. τη ρευστότητα, αλλά δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη σημασία της ρευστότητας, ούτε να θεωρήσουμε ότι είναι αυτονόητη. Όλα αυτά τα εξετάζουμε πολύ σοβαρά και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση όσον αφορά τη δημοσιονομική σταθερότητα στην ε, ζώνη του ευρώ. Βλέπουμε να υπάρχουν φούσκες, μέχρι στιγμής όχι. Βλέπουμε κάποια τοπικά φαινόμενα Περισσότερο όμως, αν όχι αποκλειστικά, ε, στην πρωτογενή αγορά ακινήτων. Σε κάποιες πόλεις βλέπουμε ότι αυξάνονται ραγδαία οι τιμές των κατοικιών, αλλά θα πρέπει να συγκρίνουμε την κατάσταση με πριν λίγο καιρό, όπου ήταν υπερβολικά χαμηλές, αδικαιολόγητα χαμηλές οι τιμές αυτές. Ε, δεν απέχουν λοιπόν, δεν έχουν αποκλίνει πολύ από, τα, από τον ιστορικό μέσο όρο και αυτό αφορά κυρίως μεγάλες πόλεις σε κάποιες χώρες. Η απάντηση λοιπόν είναι, εάν υπάρχουν ε, κίνδυνοι δημοσιονομικής σταθερότητας, ε, είναι περιορισμένοι, τοπικοί, μη συστημικοί και αφορούν συγκεκριμένες καταστάσεις. Και η απάντηση είναι ότι οι αρχές σε πολλές χώρες ε, ήδη έχουν λάβει μέτρα μακροπροληπτικού χαρακτήρα για να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Η απάντηση πάντως σίγουρα δεν είναι να αλλάξει η νομισματική πολιτική, διότι αυτό δεν θα πρέπει να είναι η ανταπόκριση σε έναν τοπικό κίνδυνο. Ευχαριστώ Μάρκ Κοβάλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις για σας. Η πρώτη αφορά μια γνώμη η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα σχετικά με το μορατόριο που θα πρέπει να ισχύσει στην περίπτωση όπου εξηγιανθεί σε εισαγωγικά μια τράπεζα όπου προβλέπεται να σταματήσει κατά κάποιο τρόπο ο χρόνος για πέντε μέρες αλλά προτείνονται ακόμα και οι καταθέσεις να δεσμευθούν προσωρινά για ένα πενθήμερο. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε λοιπόν με ποιο δικαίωμα προτείνεται να μπλοκαριστούν οι καταθέσεις των πολιτών για πέντε μέρες. Οι τρέχοντες λογαριασμοί τι σχέση έχουν. Καταλαβαίνω το τι θα πρέπει να συμβεί με τους επενδυτές, αλλά όχι με τους τρέχοντες λογαριασμούς. Και τώρα, για τα κόκκινα δάνεια. Τα διεθνή όργανα, οι διεθνείς οργανισμοί, θα πρέπει να συζητήσουν το θέμα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί μερικές φορές βλέπουμε ότι κάποια κίνητρα τα οποία δίδονται στις Ιταλικές τράπεζες δημιουργούνται διαχειριστικά προβλήματα και στην ουσία δημιουργείται μια παράλληλη αγορά στην εξαγορά ενεργών η οποία δεν είναι ιδιαίτερα υγιής. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει μια κάποια πίεση ε, σε σχέση με τα ενεργά τα οποία κατέχουν οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες και που παρουσιάζουν θα έλεγα ένα ιδιαίτερο υψηλό επίπεδο κινδύνου. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η γνώμη σας γύρω από αυτό. Κοιτάξτε, το SSM και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι δεν είναι και εδώ σήμερα συζητάμε την νομισματική πολιτική. Κοιτάξτε, εν μέρη μόνο είμαι σε θέση να συζητήσω κάποια από τα θέματα τα οποία θέσατε με πολύ γενικό τρόπο και κάποια σημεία δεν θα τα θίξω γιατί εγώ ασχολούμαι με θέματα εποπτείας και νομισματικής πολιτικής. Για το μορατόριο όμως. Η... Κρίθηκε η πρόταση αυτή θετική, γιατί σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις δημιουργείται μια κατάσταση στα πλαίσια της οποίας πρέπει να υπάρχει απαιτή ευελιξία για τη διαχείριση μιας κρίσεως. Το μορατόριο αυτό λοιπόν θα διασφαλίσει εν πολλής ότι θα υπάρξει αρκετός χρόνος για την προετοιμασία μιας θα έλεγα αξιόπιστης λύσης προλαμβάνοντας ε, ε, την χειροτέρευση των ροών ρευστότητας ε, που θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρξουν. Η εμπειρία δείχνει μέχρι τώρα ότι με τους υπάρχοντες κανόνες για μορατόριουμ σε ορισμένες χώρες δεν, δεν δείχνει η εμπειρία ότι το μορατόριουμ αυτό θα επιταχύνει τις διαλυτικές διαδικασίες. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ότι δηλαδή οι καταθέτες θα φύγουν από τις τράπεζες ακόμα πιο γρήγορα από ότι αν δεν υπήρχε το μορατόριο. Εγώ νομίζω ότι διευκολύνει μια διατεταγμένη αντιμετώπιση του προβλήματος. Βέβαια μιλάμε για ακραίες καταστάσεις πάντα να προσθέσω εδώ ότι θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω εκτιμήσεις και συζητήσεις γύρω από το θέμα του μορατόριου. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις, όπως σαν παράδειγμα η δημοσίευση μιας ξεκάθαρης και προκαθορισμένης ιεράρχησης των πιστωτών σαν εναλλακτική λύση στο μορατόριο. Να υπάρχει δηλαδή εκ των προτέρων να είναι γνωστή η ιεράρχηση των πιστωτών, έτσι ώστε η εξυγίανση να γίνεται με πιο τακτικό τρόπο από ό,τι γίνεται σήμερα. Αλλά δεν θα ήθελα ε, να μιλήσουμε μόνο για το μορατόριο, υπάρχουν και άλλα θέματα. Ταυτόχρονα, η ιεράρχηση των πιστωτών έτσι κι αλλιώς είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, ανεξάρτητα από το μορατόριο. Μιλάμε για μια τραπεζική ένωση με διαφορετικές ιεραρχίες, με άγνωστους παραμέτρους πολλές φορές. Αυτό δεν είναι τραπεζική ένωση, είναι κάτι το διαφορετικό, το ατελές. Ένα τομέα στον οποίο θα ήθελα να υπάρξει πίεση από πλευρά των πιστωτών είναι αυτός. Τώρα για τα επίπεδα, για τα χαρτοφυλάκια επίπεδου 2 και 3. Συμφωνούμε ότι τα επίπεδα 2 και 3 μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα σε κακή τιμολόγηση, σε υπερεκτίμηση και απαιτούν συνεχή εποπτική διαδικασία. Οι εποπτικές αρχές βασίζονται φυσικά στα προγράμματα τα οποία σήμερα είναι λειτουργικά και εξακολουθούν να αξιολογούν και να εκτιμούν το πώς οι τράπεζες σέβονται τους κανόνες πρόληψης, μακροπροληπτικής διαχείρισης κτλ. Οι βασικοί κανόνες είναι η αξιολόγηση περίπλοκων και σύμφετων προγραμμάτων και σε πιστοτικό επίπεδο και σε επίπεδο ομολογιών, ο έλεγχος των διαδικασιών εποπτείας, και επίσης η ανάλυση σε βάθος ε, των ε, πολιτικών ταξινόμησης που ακολουθούν τα πιστοτικά ιδρύματα. Αυτές δεν είναι οι προτεραιότητες ή δεν ήσαν οι προτεραιότητες το 2016 και το 2017 αλλά στα πλαίσια της εποπτικής διαδικασίας έχουμε στρέψει ήδη την προσοχή μας στα ενεργά, ε, στο level 3, στο επίπεδο 3. Όταν κάτι τέτοιο είναι σημαντικό για ορισμένα πιστοτικά ιδρύματα προσπαθούμε να αξιολογήσουμε σωστά τις απώλειες και τις ζημίες και με διαδικασίες εποπτείας εξωτερικές αλλά και επιτόπου εσωτερικές. Σας ευχαριστώ. Είναι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σε κάποια άλλη φάση αναλυτικότερα. είναι σαφές ε, ότι θα πρέπει να τύχουν μιας κάποια προτεραιότητας από πλευρά μα. Να πω επίσης στον κύριο Βάλλη ότι ευτυχώς το θέμα του μορατόριου είναι μια νομοθετική πρόταση. Είναι πλήρως δηλαδή στην δική μας ε, αν θέλετε διάθεση και διαχείριση. Είναι νομοθετική πρωτοβουλία. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε να είμαστε με σωστό τρόπο προσεκτικοί, δραστήριοι και επιφυλακτικοί βλέποντας τις κρίσιμες αν θέλετε πλευρές της διαδικασίας των μορατόριων. Οι διαδικασίες αυτές λόγω του αντικειμένου τους είναι πάρα πολύ περίπλοκες και απαιτούν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Άνεμανς κύριε Τράγη. Μας δώσατε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς ε, περιουσιακών στοιχείων και έτσι θα μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε. Θα πρέπει όμως να φροντίσουμε τα ωφέλη να είναι κοινά από το πρόγραμμα αυτό. Και Βέβαια είναι κάτι το οποίο αφορά την όλη μας ε, φιλοσοφία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ που εμείς δεν πιστεύουμε ότι είναι βιώσιμο. Εσείς όμως βλέπετε διαφορετικά την κατάσταση. δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, δεν είναι καθόλου βιώσιμη. Είχαμε πρόβλημα με την διερμηνία, λέει ο Πρόεδρος. U hebt er anders Η δική σας γνώμη λοιπόν είναι διαφορετική. Αναφερθήκατε στα χαμηλά επιτόκια και την προστασία του ευρώ. Δεν μπορείτε όμως να συνεχίσετε με το πρόγραμμα αυτό, διότι δεν είναι βιώσιμο. Ούτε μπορείτε να το διακόψετε. Παραμένουν λοιπόν σημαντικοί κίνδυνοι στο σύστημα. Κάτι το οποίο συζητιέται ακόμη σε ακαδημαϊκούς ε, κύκλους. Και ε, για παράδειγμα υπάρχει ο καθηγητής Κόκεν από το Άμστερνταμ που ασχολείται με τη διαχείριση του κινδύνου και λέει ότι το σύστημα αυτό είναι ευάλωτο και ότι έχουμε σημαντικότερους κινδύνους από το 2008 και δεν έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε. Επίσης, καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Χρόνικεν που εργαζόταν στην, στην Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα είπε ότι η πολιτική αυτή μόνο σε νέες κρίσεις θα οδηγήσει, νέα ύφεση δηλαδή και μόλις υπάρξει κάτι τέτοιο θα πρέπει να επιλέξουμε εργαλεία τα οποία δεν έχουμε πια στη διάθεσή μας. Μια υποθετική ερώτηση λοιπόν. Έχουμε εργαλεία στη διάθεσή μας για να αντιδράσουμε σε περίπτωση νέας ύφεσης ή νέων κλειδονισμών. The, um... Assessment on, our program, um, Όσον αφορά την αξιολόγηση του προγράμματός μας, το πρόγραμμα αυτό περιέχει από το σχεδιασμό του αρκετή ευελιξία ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σε ε, συνθήκες που αλλάζουν. Δεύτερον, όπως είπα και πριν, αυτή τη στιγμή, ενώ παρακολουθούμε προσεκτικά τους ε, κινδύνους ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εντοπίσει κινδύνους που να δικαιολογούν αλλαγές ε, στην, στην νομισματική πολιτική. Υπάρχουν τοπικοί θύλακες πιθανού κινδύνου που έχουν αντιμετωπιστεί με μακροπροληπτικά όργανα. Τούτου λεχθέντος όμως, εάν αναφέρεστε στο, πρόγραμμα που στο πρόβλημα που έχουμε συλλογικά, δηλαδή ε, την ε, έλλειψη χώρου ε, σε, σε περίπτωση κινδύνου, ναι, συμφωνώ πολύ τους μαζί σας. την έλλειψη περιθωρίου να αντιδράσουμε και εδώ σκέφτομαι κυρίως τις δημοσιονομικές πολιτικές και ας μην ξεχνάμε ότι η εμπειρία της κρίσης ε, μας έδειξε χώρες που δεν είχαν καθόλου δημοσιονομικό περιθώριο για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Τα επίπεδα χρέους, ε, τα ελλείμματά τους ήταν ήδη τόσο υψηλά που οποιαδήποτε πιθανή αύξηση θα τις αμφισβητούσαν οι αγορές. Και το είδαμε αυτό με σημαντικές συνέπειες ε, στην δημοσιονομική σταθερότητα των χωρών αυτών. Και άλλο θέμα είναι τα κρατικά ομόλογα που κατέχει το τραπεζικό σύστημα. Όποτε λοιπόν αμφισβητείται η αξιοπιστία των χωρών, βλέπουμε και μια ε, εγγενή δυναμία του τραπεζικού συστήματος. Και γι' αυτό βλέπουμε μείωση των πιστώσεων και ύφεση, όπως είδαμε στο παρελθόν. Η ανάκτηση λοιπόν περιθωρίου ε, για την άσκηση πολιτικής ε, είναι απαραίτητη. Και δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από τώρα να το κάνουμε αυτό, διότι τώρα τα πράγματα πάνε καλύτερα. Και αυτή είναι η απάντηση που έχω στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιώργος Κύρσος. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Ντράγκη, μου φαίνεται ότι ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, υφίσταται ισχυρή πολιτική πίεση μια φιλοκυβερνητική υπηρεσία η οποία εξειδικεύεται στις υποτιθέμενες ή και υπάρχουσες αν θέλετε κακού τύπου ενέργειες του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας έχει ήδη καταδικαστεί για συκοφαντική δυσφήμιση αλλά εξακολουθεί να υποστηρίζεται από την κυβέρνηση ή τουλάχιστον από σημαντικά κυβερνητικά στελέχη. Επίσης η κυβέρνηση κατηγορείται για επιλακτικές διαρροές στον τύπο στοιχείων για την Attica Bank και εδώ ο κύριος Τουρνάρας λέγει ότι δεν έχει πράξει κάτι το παράνομο. Εσείς εξακολουθείτε να θεωρείτε τον κύριο Στουρνάρα έναν έμπιστο κεντρικό τραπεζίτη και ένα έμπιστο συνεργάτη σας. Ε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια σχόλια να κάνετε για τη μεθοδολογία που ακολουθείτε εναντίον του κυρίου Στουρνάρα. Κοιτάξτε, δεν έχω συγκεκριμένα σχόλια πάνω στα θέματα αυτά να κάνω. Να πω ότι ο, ο κύριος Στουρνάρας είναι ένα έμπιστο μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έχει εργαστεί πάρα πολύ σκληρά για την ευημερία της χώρας του. If you want, you can make use of additional time on another topic. Um, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να είμαι και εγώ αισιόδοξο ε, όπω και ο πρόεδρο Δράκη για την κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ε, κατά πόσο οι συστημικές τράπεζες θα μπορέσουν να διαχειριστούν επιτυχώς ε, τα κόκκινα δάνεια. Γιατί η αξία των, ε, ε, των μετοχών πέφτει. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει καλή διαχείριση αυτής της κρίσης των κόκκινων δανείων ή πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει επιπλέον πρωτοβουλία για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτές τις ε, δυσκολίες ε, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, έχω σχολιάσει και στο παρελθόν ε, την κεφαλαιακή κατάσταση των τραπεζών σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όμως τα κόκκινα δάνεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. η απόφαση να μην υπάρξει ηλεκτρονική και φυσική ε, δημοπράτηση μέχρι το τέλος της χρονιάς, αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Α, άλλαξε αυτή η απόφαση. Α, τότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό, καλός είναι γεγονός ε, ότι η διάθεση των κοκκίνων, των κόκκινων δανείων είναι πράγματι ένα πολύ δύσκολο ε, πρόβλημα και πρέπει οι, οι κοινωνικές πτυχές όλης αυτής της διαδικασίας ε, να καλυφθούν και όντως να ληφθούν υπόψη από την ε, κυβέρνηση. Και όντως αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα γίνει ένα τεστ αντοχής για τις ελληνικές τράπεζες νωρίτερα από ό,τι για τις ε, άλλες τράπεζες. Ε, γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα των κόκκινων δανείων πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικότητα και γνωρίζουμε, όπως είπα και προηγουμένως, ότι η κατάσταση, οι συνθήκες χρηματοδότησης δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί. Θα έχουμε όμως, νομίζω, μια καλύτερη εικόνα του πώς έχουν τα πράγματα με ε, το τεστ αντοχής που θα γίνει νωρίτερα για τις ελληνικές τράπεζες ε, και θα ξέρουμε τότε αν πρέπει να υπάρξει κάποια ε, διορθωτική δράση και αν υπάρξει αυτή η ανάγκη θα γίνει πριν από το τέλος της αξιολόγησης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, Φερνάντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι μέχρι τώρα λάβατε αρκετές και σημαντικές ερωτήσεις και δώσατε αρκετές απαντήσεις που ξεκαθαρίζουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στα πλαίσια των διαδικασιών ανάκαμψης της ζώνης ευρώ που είναι σαφής πλέον θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται με το κενό παραγωγής το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί και σε ποιο βαθμό ο πληθωρισμός θα μπορούσε εν μέρη να οφείλεται και στην πορεία των τιμών της ενέργειας και να φτάσει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το 2%. Θα θέλαμε λοιπόν να μας δώσετε λίγο πιο αναλυτικά τις προοπτικές της ζώνης ευρώ σε σχέση με τα θέματα αυτά. Τώρα, η συζήτηση η οποία γίνεται σε σχέση με την έννοια της σταθερότητας των τιμών. Είναι μια ακαδημαϊκή λίγο συζήτηση. Δεν ξέρω αν το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, μπορεί να θέσει σε κάποια φάση υπό αμφισβήτηση το 2% αλλά θα ήθελα να γίνει μια, περισ... μια συζήτηση σαν και αυτή η οποία γίνεται σε ακαδημαϊκό επίπεδο για τη λεγόμενη νομισματική πολιτική για το ποιος είναι ο ρόλος ε, του δημογραφικού παράγοντα που επηρεάζει τις αναπτυγμένες οικονομίες και την εφαρμοσμένη πλέον νομισματική πολιτική. και μήπως θα πρέπει να μην τεθεί στόχος μόνο σε σχέση με τον πληθωρισμό αλλά να τεθεί σε σχέση με την σταθερότητα των τιμών. Και αυτό το 2% το οποίο συζητιέται σήμερα είναι κάτι το σχετικά συμμετρικό διότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι μπορεί να συμβαίνει και η ερμηνεία για το 2% είναι κάτι το πάρα πολύ σχετικό και ο καθένας μπορεί να θεωρήσει ότι είναι και στα, στα όρια κάποιου λάθους. Θα πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουμε τους στόχους ε, της νομισματικής πολιτικής που δεν είναι αποκλειστικά το θέμα των τιμών, είναι φυσικά και το θέμα της αγοράς ακινήτων και να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να βασιστούμε σε αυτούς όπως το ύψος του ΑΕΠ και τα λοιπά. Ίσως μια συζήτηση θεωρητική αλλά θα θέλαμε περισσότερα στοιχεία γύρω από όλα αυτά. Δεν έχουμε συζητήσει εμείς κάποιες πιθανές αλλαγές στους ορισμούς που δίνουμε στη σταθερότητα των τιμών και υπάρχουν κάποιοι λόγοι επαρκής γι' αυτό. Καταρχάς δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο ή τουλάχιστον στις ε, μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες στον κόσμο έχουν υιοθετήσει τον ορισμό που χρησιμοποιούμε σήμερα για τη σταθερότητα των τιμών στα τέλη της δεκαετίας του 90 μετά από εμπειρίες που υπήρχαν και ιδιαίτερα στην Ιαπωνία. Και νομίζω ότι η αιτιολόγηση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν συζητάμε το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο ένας από αυτούς έχει σχέση με αυτό που θα ονόμαζα αξιοπιστία. Για να αλλάξει κανείς τον στόχο αυτή τη στιγμή δεν έχει σε σχέση να το πετύχει το στόχο αυτό δεν είναι δείγμα αξιοπιστίας. Αν θα επιλέγαμε ένα διαφορετικό στόχο τότε θα μας κατηγορούσαν ότι έχει ανέβει πάρα πολύ ο πληθωρισμός, ότι θα πρέπει να αλλάξουμε ακόμα μία φορά και να υιοθετήσουμε σαν κεντρικό στόχο ένα χαμηλότερο πληθωριστικό επίπεδο. Συνεπώς λοιπόν δεν είναι σωστή η στιγμή για να θέσουμε σε αμφισβήτηση τους ορισμούς αυτούς. Επιπλέον θα πω ότι το επίπεδο των προσδοκιών σταθμίζεται και εξαρτάται από τους ορισμούς αυτούς. Το να συζητήσουμε λοιπόν κάποιες πιθανές αλλαγές στους ορισμούς είναι κάτι το οποίο θα λειτουργούσε αποσταθεροποιητικά και προς τις δύο κατευθύνσεις. Συνεπώς λοιπόν τέτοιου είδους συζητήσεις για αλλαγές ορισμών στον τομέα της σταθερότητας των τιμών δεν είναι χρήσιμες. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην επίτευξη των στόχων. Αυτό κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι ο καθοριστικός στόχος της εντολής μας. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε Ντράγκη ε, που ήρθατε να μας συναντήσετε σήμερα για αυτή την ανταλλαγή απόψεων ε, η οποία, η οποία πάντοτε είναι πολύ χρήσιμη και πολύ απεικοδομητική. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά την κρίση ε, υπό την ηγεσία σας αλλά και του προκατόχου σας του κυρίου Τρισέ είχε αποφασιστική δράση για τη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Ε, ανακοινώθηκε και επανέρχομαι σε κάτι που το έχετε ξαναπεί αλλά ίσως ενδεχομένως να μπορείτε να μας δώσετε κάποια συμπληρωματικά στοιχεία είχε ανακοινωθεί μία μείωση ε, του προγράμματος ε, αγορών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα ήθελα να μάθω ποιοι είναι οι κίνδυνοι κατά τη γνώμη σας ακόμη και αν οι πρώτες ενδείξεις το γεγονός ότι δεν υπήρξαν αντιδράσεις από τις αγορές είναι μάλλον θετικό εσείς ε, ανοιχνεύετε κινδύνους και θα ήθελα συγκεκριμένα να μάθω ποιος θεωρείται ότι θα είναι ο αντίκτυπος ε, στην ευρωπαϊκή οικονομία και ειδικότερα στι τράπεζες, ε, δεδομένου ότι εκείνε κυρίω χρηματοδοτούν την οικονομία. Έχω και μία δεύτερη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, που αφορά την νομισματική πολιτική των άλλων υπερδυνάμεων, όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ιαπωνία, η Κίνα και θα ήθελα να μου πείτε πώς λαμβάνετε υπόψη τον αντίκτυπο το δικό τους ε, στην ευρωπαϊκή οικονομία όταν παίρνετε τις δικές σας αποφάσεις ε, νομισματικής πολιτικής. Και αν έχω κάποια δευτερόλεπτα ακόμη στη διάθεσή μου, μία τρίτη ερώτηση θα ήθελα να σας θέσω. Για τη γύρανση του πληθυσμού. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πώς μπορούμε να συνδυάσουμε ε, επιτόκια τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας όπως επίσης ε, και την αποταμίευση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της γύρανσης του πληθυσμού. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ. Όπως είπατε κι εσείς, ε, οι αποφάσεις μας ε, επικροτήθηκαν με μία αντίδραση από τις αγορές, που είναι πάντοτε η ε, καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ε, κάτι το οποίο δείχνει ότι η προσεκτική διαμόρφωση των, στοιχείων της νομισματικής πολιτικής μας όπως είναι οι μηνιαίες ροές, η απόφαση να συνεχίσουμε ε, τις επανεπενδύσεις των πληρωμών των ληξιπρόθεσμων ε, χρεογράφων όπως επίσης οι γραμμές μας για τα επιτόκια και το MRO όλα αυτά τα στοιχεία είναι τμήμα μία μιας ε, σύνθετης αρχιτεκτονικής μέσων που βέβαια αντικατοπτρίζουν την ε, γενικότερη βελτίωση της κατάστασης ε, και της, της κατάστασης της οικονομίας και της Ευρωζώνης. Αυτή τη στιγμή, επειδή με ρωτήσατε ποιος είναι ο κίνδυνος που προβλέπουμε, αυτή τη στιγμή ένας από τους κινδύνους που διαβλέπουμε είναι η μη επιθυμητή, ο μη περιορισμό περιορισμός της ε, οικονομικής πολιτικής που μπορεί να προέρχεται από εξωτερικούς παράγοντες, θα μπορούσε κανείς κάποιο να σκεφτεί καταστάσεις σε άλλα μέρη του κόσμου που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ε, κάτι τέτοιο από τον γεωπολιτικό κίνδυνο μέχρι το ε, γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσαρέσκειες όσον αφορά την, ε, τα προγράμματα άλλων ε, χωρών. Αυτό μπορεί να είχε ως αποτέλεσμα προσδοκίες που αυτή τη στιγμή έχουν τιμολογηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θα χρειαστεί δηλαδή μία διόρθωση της αγοράς που μπορεί να ε, οδηγήσει σε ε, περιορισμό ε, της χρηματοδότησης και των συνθήκων χρηματοδότησης στην Ευρωζώνη. Και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Πάντοτε το έχουμε αυτό στο μυαλό μας ως πιθανότητα. Και να απαντήσω έτσι και στη δεύτερη ερώτησή σας αν λαμβάνουμε υπόψη την, τι γίνεται με την νομισματική πολιτική και ποιος είναι ο αντίκτυπος νομιματικής πολιτικής άλλων χωρών του κόσμου, ε, η σταθερότητα των τιμών ε, ορίζεται ε, σε επίπεδο ευρωζώνης, όμως σε άλλες χώρες τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μπορεί να υπάρχει μια διτή ένας διτός ορισμός τιμών. Αυτό που προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη εμείς στις πληροφορίες μας είναι νομισματικές πολιτικές άλλων χωρών. Όμως στην περίπτωση μεγάλων οικονομιών, όπως είναι η Ευρωζώνη για παράδειγμα, εμείς ουσιαστικά έχουμε ως γνώμονα τις δικές μας εσωτερικές, τη δική μας εσωτερική κατάσταση. Εντάξει, βεβαίω ε, κοιτάζουμε τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίο όμω είναι διαφορετικό από το δικό μα. Ε, προσπαθούμε να παραμένουμε αρκετά ε, ανοιχτοί, χωρί όμω να θεωρούμε ότι είμαστε μια μικρή οικονομία που θα υποφέρει. Είμαστε αρκετά μεγάλοι ως ευρωζώνη, ώστε οι συνθήκες που υπάρχουν να είναι αρκετά κυρίαρχες σε σχέση με τον αντίκτυπο που μπορεί να προέλθει από ε, προβλήματα σε άλλες μεγάλες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πέντρο Σίλβα Μπερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Τράγη, δεν υπάρχει αμφιβολία νομίζω ότι η νομισματική πολιτική έχει παίξει ρόλο κλειδί στην οικονομική ανάπτυξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, έλαβε για άλλη μια φορά πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επικροτώ την αναπροσαρμογή των εργαλείων της ε, νομισματικής πολιτικής, ε, διότι θέλουν να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο οικονομικών κινήτρων και βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και βιώσιμο επίπεδο του πληθωρισμού. Συνήθως ο κόσμος κοιτάει τους μεγάλους τίτλους. Ε, τα επιτόκια θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα και μάλιστα μετά το τέλος ε, του προγράμματος ε, αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Το πρόγραμμα αυτό θα διατηρηθεί μέχρι να έχουμε αποδεκτά επίπεδα πληθωρισμού και προβλέπονται οι αγορές σε 30 δισεκατομμυρίων ευρώ το μήνα ε, το 2018. Περιμένουμε λοιπόν ε, σημαντικά οικονομικά κίνητρα. Θα ήθελα όμως να επικεντρωθώ στον ξεχασμένο πυλώνα της ε, νομισματικής πολιτικής. Η ανακοίνωση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα επανεπενδύσει όλες τις πληρωμές από αξιόγραφα που λήγουν για όσο αυτό είναι απαραίτητο. Νομίζω ότι αυτό είναι υψίστης σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και θα ήθελα να ε, αναπτύξω τις ε, συνέπειες αυτού του μέτρου. Είπατε ότι αυτό θα είναι ευνοϊκό για τη ρευστότητα. Θα διασφαλίσει και την ε, σωστή νομισματική πολιτική. Αυτό το μέτρο μπορούμε να περιμένουμε να, ότι θα συμβάλλει και σε πιο ισορροπημένη κατανομή των κινήτρων σε όλη την Ευρωζώνη. Όλοι ξέρουμε ότι οι αγορές ανακράτος μέλος ε, περιορίζονται ε, από τις ε, απαιτήσει σχετικά με τα κεφάλαια και αυτό σημαίνει ότι αγορές η κάποια κράτη-μέλη είναι περιορισμένες, όπως είναι η Πορτογαλία. Τα ποσά από αξιόγραφα που λήγουν θα επανεπενδυθούν. Αυτό σημαίνει ότι χώρες όπως η Πορτογαλία μπορεί να περιμένει υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Μας ε, περιορίζει η κλίδα κατανομής ε, κεφαλαίων και οι αρχές μας. Όσον αφορά όμως τη σύγκληση μεταξύ των χωρών των, της Ευρωζώνης, ήδη έχουμε διαπιστώσει σημαντικό βαθμό σύγκλησης ε, σύμφωνα με μια σειρά μέτρων. Στην εισαγωγή μου ανέφερα την ε, ανάπτυξη και την προστιθέμενη αξία. Και βλέπουμε θετικές εξελίξεις σε, σε χώρες της Ευρωζώνης. Ε, διαπιστώσαμε ότι... διαπιστώσαμε επίπεδα του ύψους του 1997. Βλέπουμε λοιπόν ε, σύγκληση με μεγαλύτερη ανάπτυξη σε χώρες που είχαν χαμηλή ανάπτυξη. Με την έννοια αυτή λοιπόν ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα και περιμένουμε αυτή η πορεία να συνεχιστεί. Αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες ειδήσει της ανάκαμψης. Ότι δεν είναι πια τοπικό φαινόμενο, είναι ευρύτερο φαινόμενο της Ευρωζώνης. Όσον αφορά το πρόγραμμα επενδύσεων, δημοσιεύουμε ε, την ε, τιμή για κάθε ε, αξιόγραφο που λύγει για το επόμενο 12 μήνο και αυτά τα ποσά εξαγοράς ε, θα ανέλθουν σε 11 δισεκατομμύρια κατά μέσο όρο ανά μήνα, αν και μπορεί να υπάρχουν σημαντικέ διαφορές από μήνα σε μήνα. Διότι είπαμε ότι η επαναγορές γενικά θα γίνονται με τη λήξη τους. Αλλά για να έχουμε αρκετή ευελιξία και να αποφύγουμε ανεπιθύμητες συνέπειες, αυτές οι επαναγορές μπορούν να γίνουν μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Θα υπάρξουν λοιπόν διαφορές. Αυτές οι επανεπενδύσεις θα γίνουν εγκαίρως, όπως είπα, και θα πραγματοποιηθούν εντός των ίδιων ε, ε, δικαιοδοσιών ε, με τις αρχι με τα αρχικά αξιόγραφα, διότι θέλουμε να ακολουθήσουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν την κλίδα κατανομής κεφαλαίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Πρόεδρε που ήρθατε εδώ. Ερώτηση σχετικά με την νομισματική πολιτική να πω καταρχάς ότι νομίζω ότι ήσασταν πολύ μετριόφρονε κατά την περιγραφή της κατάστασης στην Ευρωζώνη. Εμένα μου φαίνεται ότι τα στοιχεία δείχνουν ε, όχι μόνο βελτίωση σε σχέση με προηγούμενα έτη, αλλά ουσιαστικές αλλαγές. Η αύξηση του ΑΕΠ από το 2013 έχει αυξηθεί σημαντικά. Το 2016 βλέπουμε μείωση συνεχή της ανεργίας από το 2013 βλέπουμε να μειώνεται επίσης η μακροπρόθεσμη ανεργία, η ανεργία μακράς διαρκείας, ε, αλλά και ο πληθωρισμός ε, βρίσκεται κοντά στο μηδέν. Ε, νομίζω όμως ότι θα αρχίσουν να βελτιώνονται και οι μισθοί. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε βελτιώσεις, διότι η οικονομία φαίνεται να είναι στεναρή. Καταλαβαίνω ότι τονίζετε την ποσοτική πλευρά της νομισματικής πολιτικής ε, και λέτε ότι ε, έχουμε ένα σημαντικό ε, κενό, αρνητική παραγωγή, το οποίο θα πρέπει να κλείσει ε, η οικονομική ανάκαμψη όμως πιστεύω ότι θα επιταχυνθεί και ότι σύντομα θα επιφέρει βελτιώσεις σε πολύ σημαντικούς τομείς όπως είναι η απασχόληση και οι αμοιβέ. Ε, όλα αυτά με πολύ χαμηλά επιτόκια ονομαστικά τουλάχιστον. Ε, και η δεύτερη μου ερώτηση πώς ε, συνδυάζονται τα πολύ χαμηλά επιτόκια με την ποσοτική σας πολιτική. Δεν αποτελεί επιλογή το να αυξηθούν τα επιτόκια διατηρώντας την ποσοτική σας πολιτική ως έχει ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ε, της ε, ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τη θετική σας εκτίμηση σχετικά με την ε, ανάκαμψη της Ευρωζώνης και είμαστε πεπισμένοι ότι θα δούμε αλλαγές στους ονομαστικούς μισθούς που θα οδηγήσουν σε πιο πιστική ανωδική τάση τον ονομαστικό πληθωρισμό από ό,τι είδαμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα είχαμε πολύ ελαφρές ε, τροποποιήσεις τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Δεν είδαμε όμως μια απιστική ανωδική τάση. Και ο λόγος είναι αυτός που αναφέρατε. το ότι δεν είδαμε σημαντικές αυξήσεις στους ονομαστικούς μισθούς. Από την άλλη, Εξετάζοντας τις ε, βελτιώσεις ε, στο, ε, αρνητικό κενό, στο κενό παραγωγής, Βλέπουμε ακριβώς αυτήν την διτή πραγματικότητα. Από τη μία πολύ ε, πιστικές εξελίξεις όσον αφορά την απασχόληση. τη, βλέπουμε επίσης ισχυρή κατανάλωση, επενδύσεις που συνήθως ε, ήταν το ε, ε, χαμηλότερο τμήμα, ο χαμηλότερος τομέας στην ανάκαμψη τώρα ανέρχεται σε 45%. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι οι παράγοντες που οδηγούν σε ανάκαμψη μας δείχνουν ότι όχι μόνο τα επίπεδα αλλά και η τάση αυτής της ανάκαμψης θα συνεχιστεί Ε, με τον ίδιο τρόπο, αν όχι ε, ακόμα πιο ανωδικά από ό,τι στο παρελθόν. Από την άλλη, είμαστε υπομονετικοί και ε, ακριβείς στον υπολογισμό των κινήτρων για βελτίωση των οικονομικών συνθήκων. στο πλαίσιο αυτό έχουμε συζητήσει επανειλημμένα ακριβώ αυτό που λέτε εσείς. Την ε, σειρά δηλαδή των μέτρων μας, ξεκινώντας από πέρσι, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και ε, η ακολουθία αυτών των μέτρων είναι σημαντική. Γι' αυτό τα επιτόκια θα παραμείνουν στα παρόντα επίπεδα για αρκετό διάστημα μετά τη λήξη του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι έτσι οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων ελέγχεται. Και η καμπή απόδοσής μας σε σχέση με άλλες δικαιοδοσίες ε, έχει παραμείνει καλή, ε, όπως επίσης ε, και οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις λόγω του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ιάκοπ Φονβάιτσεκ. Thank you, Chair. Um, President Draghi, um, of course we're extremely grateful. Φυσικά και είμαστε ευγνώμονες για τον, για τον τρόπο με τον οποίο η νομισματική πολιτική έχει βοηθήσει τα τελευταία χρόνια και μας έχει οδηγήσει στην κατάσταση την οποία έχουμε μπροστά μας σήμερα. Ταυτόχρονα έχω την αίσθηση ότι η επιφυλακτικότητα την οποία επιδεικνύεται ότι στα πλαίσια μιας εύθραυστης κατάστασης δεν θα πρέπει να πιέσουμε πολύ είναι κάτι το σωστό. Θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα όμως για τη νέα κανονική κατάσταση αν θέλετε. Υπάρχουν κάποιες προσδοκίες τις οποίες θα πρέπει να καλύψουμε. Υπάρχει βέβαια η αγορά εργασίας η οποία δεν δείχνει ακόμα κάποια στοιχεία αλλά η νέα κανονική κατάσταση θα είναι τέτοια έτσι ώστε τα επιτόκια θα εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ χαμηλά και σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης και εφόσον οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμείνουν στα επίπεδα τα οποία έχουμε σήμερα ε, δεν είναι σαφές αν θα κινηθούμε δεξιά ή αριστερά του χρυσού κανόνα. Κάτι το οποίο από μόνο του δημιουργεί μια νέα εύθραυστη κατάσταση για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Μήπως θα πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο στα πλαίσια του νέου παραδείγματος θα διατηρήσουμε την ισορροπία. Και δεύτερον, η βασική πρόκληση για σας ως κεντρικός τραπεζίτης. Με ποιο τρόπο θα μπορέσετε εσείς να ασκήσετε μια νομισματική πολιτική στα πλαίσια αυτής της νέας κατάστασης όταν ε, το περιθώριο κίνησης είναι πάρα πολύ περιορισμένο και δεν μιλάμε για τους ε, επόμενους μήνες κάποιες δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν, ο χώρος μέσα στον οποίο μπορείτε να κινηθείτε πολιτικά είναι πάρα πολύ περιορισμένος, είναι συρρυκνωμένος. Οπότε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε ακριβώς αυτόν τον νέο κανόνα, τον τόσο εύθραυστο όμως. Σας ευχαριστώ. Η παρούσα κατάσταση είναι μια κατάσταση συνεχούς βελτίωσης και στα πλαίσια της ανάπτυξης του ΑΕΠ και βελτίωσης της αγοράς εργασίας. Αυτό τώρα θα οδηγήσει σε μια νέα κατάσταση όπου τα επιτόκια θα εξακολουθούσε να είναι, τα πραγματικά επιτόκια θα πρέπει να είναι πάντα πολύ χαμηλά. Νομίζω ότι η κατάσταση εξελίσσεται συνεχώς και με τρόπο διαφορετικό από τον υπόλοιπο κόσμο. Η ρυθμή ανάπτυξή μας είναι υψηλότερη από ό,τι στο παρελθόν. Βλέποντας τα παλαιά στοιχεία για τις δυνατότητες της αναπτυξιακές, έχουμε ξεπεράσει τους μέσους όρους εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε ποια θα είναι η νέα κανονική κατάσταση, οι νέοι κανόνες για την Ευρωζώνη. Δεν μπορώ να πω. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι εσείς ε, αυτό το οποίο προτείνετε, το συμπέρασμα στο οποίο και το αναφέρατε και αυτό, είναι ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα θα καταστεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτής της νέας κανονικής κατάστασης. Και να πω εδώ ότι αρκετά μέτρα έχουν ήδη ληφθεί στον τομέα αυτό και θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής που θα ακολουθηθεί έτσι ώστε τα εύθραυστα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει η νέα κατάσταση να μην γίνουν πραγματικότητα σε επίπεδο που θα μπορούσε να διαταράξει το περιβάλλον μέσα στο οποίο πράγματι τα επιτόκια θα συνεχίσουν να είναι στα επίπεδα που είναι σήμερα. Μια τέτοια κατάσταση με καλύπτει εμένα η αγορά εργασίας να βελτιώνεται, οι ρυθμοί ανάπτυξης να είναι ψηλοί και τα επιτόκια χαμηλά. Είναι όμως σαφές ότι στα πλαίσια μιας τέτοια κατάσταση και οι μακροπροληπτικές και οι μικροπροληπτικές πολιτικές έχουν μεγάλη σημασία. Γιατί πράγματι ο χώρος για τις μακροπρόθεσμες πολιτικές, όπως είπατε, είναι περιορισμένη. Και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο ισχύουν αυτά που είπα προηγουμένως. Ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την παρούσα συγκυρία έτσι ώστε να αναδημιουργήσουμε τον απαιτούμενο χώρο για την δημοσιονομική μας ε, πολιτική σε επίπεδο διαφθρωτικό. Ο καλύτερος τρόπος ε, να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα κανονική κατάσταση είναι να διαμορφώσουμε χώρο κίνησης και από την άλλη στα πλαίσια των μακροπροληπτικών πολιτικών να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν διαταράξεις της εξελικτικής αυτής διαδικασίας. Σας ευχαριστώ. Μουρεσάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω για το CSPP και για την επικοινωνία των ε, ε, αποφάσεων νομισματικής πολιτικής. Θα ήθελα για την πρώτη μου ερώτηση να σας πω αν έχετε αλλάξει τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το CSPP ε, και αν το CSPP σταδιακά καταργηθεί στο μέλλον, μήπως υπάρξει και πάλι ανάγκη ε, να καταστεί και πάλι απαραίτητο και τότε ε, τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα ε, αναπροσαρμοστούν αν χρειαστεί να ξαναυπάρξει ένα GSPP στο μέλλον. Και όσον αφορά την επικοινωνία γύρω από την νομισματική πολιτική, είχατε πάει την περασμένη εβδομάδα ε, με τον ε, πρόεδρο της, ε, της Ιαπωνικής Τράπεζας σε μια υψηλού επίπεδου επικοινωνία διάσκεψη για την επικοινωνία για τα θέματα αυτά. Εσείς πώς θεωρείτε ότι μπορείτε να βελτιώσετε την επικοινωνία δεδομένου ότι πρέπει οι κεντρικές τράπεζες να μπορούν να εξηγούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις δικές τους χώρες. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ αυτής της ε, ε, ε, επισήμανσης σε επίπεδο εθνικό αλλά και με το γεγονός ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες κατακρίνουν συχνά ε, την επικοινωνία αυτή. Ε, ναι, για το πρώτο σας ερώτημα, εμείς ε, πιστεύουμε ότι τα προγράμματα αγοράς, των τριών, τα τρία προγράμματα για το ιδιωτικό τομέα, το CSPP, το ABSPP και το πρόγραμμα Cover Bonds υπαριθμών 3, Θεωρούμε ότι ε, θα εξακολουθούν να ε, παραμένουν ε, και αρκετά εκτεταμένα το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει σε αλλαγές των συνθήκων των αγορών μέσω της αναδιανομής των όγκων αγορών μεταξύ των τεσσάρων προγραμμάτων. Οπότε τέτοια αναδιανομή έχει γίνει στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν ε, ήταν περιορισμένη εμβέλεια αυτές, ε, αυτή η αναδιανομή αναμένεται να συνεχιστεί. Όσον αφορά λοιπόν την αναδιανομή, εμείς θεωρούμε ότι θα εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς και το PSBB ε, λειτουργεί στην, πιο, στην αγορά με την μεγαλύτερη ρευστότητα και σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάσει τη διακύμανση ε, των αγορών στοιχείων ε, και άλλων προγραμμάτων. Όσον αφορά τώρα το, τη νομισματική πολιτική και την επικοινωνία αυτής, η διάσκεψη αυτή ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα, καταρχάς γιατί ε, έδειξε τη σημασία ε, του πόσο σημαντική τη σημασία της επικοινωνίας, της νομισματικής πολιτικής, αλλά αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε φορά. Όσο σαφέστερη είναι η επικοινωνία μας, τόσο καλύτερα γίνεται κατανοητή από τις αγορές. Η ίδια επικοινωνία είναι ένα μέσο νομισματικής πολιτικής η ίδια. Οι κατευθυντήριες γραμμές... Ε, ε, ως μέσο επικοινωνίας έχουν αποτελέσει ένα πολύ πιο αποτελεσματικό εργαλείο επικοινωνίας ε, ε, όπως ανακοινώσεις της τράπεζας στο παρελθόν. Γι' αυτό λοιπόν έχει νόημα η αυξημένη προσοχή στην επικοινωνία. Είναι ανα, αναπόσπαστο τμήμα της νομισματικής μας πολιτικής αλλά και της λογοδοσίας μας. Η λογοδοσία είναι σημαντική γιατί είμαστε ανεξάρτητοι και είμαστε είμαστε ανεξάρτητοι στο πλαίσιο μίας εντολής. Οπότε ε, πρέπει να λογοδοτήσουμε και ε, στη διάσκεψη αυτή άκουσα ε, μια τέτοια παρέμβαση ε, πρέπει να πω ότι είμαστε ανεξάρτητοι, ε, αλλά αυτό αποφασίζεται από τους ε, ερετούς εκπροσώπους. Εμείς δεν εκλεγόμαστε από κανέναν, οπότε αξιολογούμαστε βάσει της λογοδοσίας μας. Είναι λοιπόν η λογοδοσία μας ένα πάρα πολύ σημαντικό καθήκον, γιατί αυτό είναι ο έλεγχος που μας γίνεται και η επικοινωνία μέσω της λογοδοσίας γίνεται ένα μέσο νομισματικής πολιτικής. Και είπα μάλιστα ότι ε, οι υποθέσεις του ε, δικαστηρίου μας επέτρεψαν να δούμε πόσο καλά συμμορφωνόμαστε με την εντολή μας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο έλεγχος της συμμόρφωσής μας. Είναι ε, διτός ο ρόλος λοιπόν. Είναι υποχρέωσή μας, αλλά είναι και μέσο νομισματικής πολιτικής πλέον. Υπερβώς ε, ευχαριστώ πολύ. Σα είπα στο πρώτο μου ερώτημα, στην πρώτη μου ερώτηση, ότι δεν θα σας έκανα ερώτηση σε σχέση για την μείωση των κινδύνων στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωση. Θα το κάνω όμως, γιατί ε, επειδή άκουσα την ανταλλαγή απόψεων ω τώρα, εγώ πιστεύω ότι το θέμα του ντι ε, έχει αναφερθεί από εδώ και από εκεί και ο καθένας θεωρεί ότι όλοι θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ε, μην ε, παραμείνει ε, ε, μπλοκαρισμένο, πρέπει να ξεμπλοκάρει, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη ε, στο τραπεζικό σύστημα και αν δεν μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε αυτό το σύστημα, τότε θα μπλοκάρουν και άλλα θέματα που σχετίζονται με αυτό. Δύο στοιχεία λοιπόν θα ήθελα να ε, θέσω και να επιμείνω σε αυτά. Κρίμα που η κυρία Αγγεν δεν είναι εδώ, αλλά ενδεχομένω να, να την ενημερώσουν. Πάντα μιλάμε για τη μείωση κινδύνων και την κατανομή κινδύνων. Όμω, να σα πω την αλήθεια, ε, κάθε φορά τη μείωση κινδύνων ε, μας την αναφέρεται σε κάθε ανταλλαγή απόψεων στο, πλαίσιο διαλόγου αυτού και εξακολουθούν να υπάρχουν. Ε, ε, πού έχει αυξηθεί λοιπόν η κατανομή των κινδύνων, ε, δηλαδή αρχίζει να υπάρχει μία τάση Υπάρχει ένας παραλληλισμός μεταξύ των δύο, αλλά πάντοτε υπάρχει μείωση κινδύνων ε, και αναδιανομή και διανομή των κινδύνων. Ε, δεν είναι δυνατόν το ένα να έρχεται σε αντίθεση με το άλλο. Ε, είπατε fully fledged issuance. Τι, ποιο είναι το, το κρίσιμο σημείο. Η ιδέα είναι ότι πρέπει να θέσουμε όρους για το πέρασμα από τη μία φάση στην άλλη βάσει της προόδου των διαπραγματεύσεων ή πρέπει να κοιτάμε τον τελικό στόχο, δηλαδή πού θέλουμε να βρισκόμαστε στο τέλος και να βρούμε έναν τρόπο να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτω με το τελευταίο που είπατε. Όντω πρέπει να έχουμε έναν κοινό συμπεφωνημένο στόχο και ε, πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να φτάσουμε εκεί. Και αν δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία στην ε, κατανομή του κινδύνου, ε, δεν ε, είχα τέτοια πρόθεση. Είναι προφανώ ότι αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να συνάδουν, είναι προφανέ. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένα ταξίδι. Είναι ένα ταξίδι που το κάνουμε μαζί, ε, κατανομή κινδύνου και μείωση κινδύνου πρέπει να συμβαδίζουν. Ο τρόπο λοιπόν να κάνουμε αυτό το ταξίδι παρουσιάζεται στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι που να είναι ταχύτεροι ή βραδύτεροι. Εξαρτάται. Το σημαντικό όμω είναι να μπορούμε να συμφωνούμε επί του τελικού και δεν το, δεν το έχουμε συμφωνήσει αυτό. Δεν υπάρχει αυτός ο κοινό στόχος ε, που να τον έχουμε συμφωνήσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Και το δεύτερο είναι πώς θα φτάσουμε σε αυτόν τον τελικό στόχο. Το γεγονός ότι αυτό το ταξίδι είναι ε, σαφώς ε, καθορισμένο επειδή ανέφερε και τη λογοδοσία προηγουμένως, είναι, είναι, είναι ένα ταξίδι ε, για το οποίο πρέπει να υπάρχει λογοδοσία, να ξέρουμε τι γίνεται σε κάθε φάση του ταξιδιού και τι θα έπρεπε να γίνει. Εγώ έτσι βλέπω αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μουρεσάν. Κοιτάξτε, δεν θέλω να πάρω το λόγο επειδή κάνω τι ε, διαπραγματεύσει του προπολογισμού, αλλά επειδή ο συνάδελφο έπρεπε να φύγει, μάλλον είναι άρρωστο σήμερα και δεν μπόρεσε να κάνει την ερώτησή του και θα ήθελε να τη θέσει μέσω εμού. Πρώτον, όσον αφορά τα κέρδη τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ε, η ομάδα εργασία ιδίων πόρων ε, υψηλού επίπεδου υπό την ηγεσία του Μάριου Μόντι μιλά για την ε, χρηματοδότηση και τη νέα χρηματοδότηση ιδίων πόρων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης και το ερώτημα βέβαια είναι ποια είναι η δική σας άποψη ως προς αυτό και αν θεωρείτε ότι είναι ένας κίνδυνος για την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζης κατά πόσο, ε, αν δηλαδή... Ε, ε, ε, ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία και το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το ψηφιακό νόμισμα. Ε, κατά τα τελευταία χρόνια ε, έχουν εμφανιστεί πολλά ε, τέτοια ε, νομίσματα και αυτό θα έχει αντίκτυπο βέβαια στο μονοπόλιο των κεντρικών τραπεζών για την έκδοση χρήματος και τη δυνατότητα ελέγχου της παροχής χρήματος και το ερώτημα του συναδέλφου είναι κατά πόσο πιστεύετε ότι αυτού του είδους τα νομίσματα μπορούν να διακινδυνεύσουν αυτό το μονοπόλιο των κεντρικών τραπεζών και αν υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι γύρω από αυτήν την εξέλιξη των ψηφιακών νομισμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Για το πρώτο σας ε, ερώτημα, ε, η εκχώρηση ε, των, ε, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η, των κερδών στον ενωσιακό προϋπολογισμό αντίθετα με το ότι όσα είπαν κάποιοι, δεν, δεν αντιτίθεται στην πολιτική των οικονομικών αποθεμάτων ε, βάσει του άρθρου 23α. Αλλάζει τον αποδέκτη ε, των ε, κερδών και αυτή η αλλαγή θα σήμαινε αλλαγή του κανονισμού άρθρο 33 ένα αλφα που θα έπρεπε να αλλάξει, που διέπει την ε, κατανομή ε, των ε, υπολοιπωμένων κερδών μετά την, το κλείσιμο του ισολογισμού κέρδους και απολειών. Όταν βλέπουμε όμως ε, το πόσο χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, ποιοι είναι οι χρήστες, ποιος είναι ο αντίκτυπος ε, της χρήσης του στην πραγματική οικονομία, ε, πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι ακόμη για την ώρα πολύ περιορισμένα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για τις κεντρικές τράπεζες. Γενικότερα όμως οι ψηφιακές τεχνολογίες και άλλες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είναι ε, μία εξέλιξη την οποία θα έπρεπε να βλέπουν ε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι κεντρικές τράπεζες αλλά και οι επόπτες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πολλές κεντρικές ε, τράπεζες των ε, κρατών μελών ήδη το επεξεργάζονται εδώ και πολλούς μήνες και μπορούμε να κάνουμε έναν συντονισμό στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και άλλες ενέργειες έχουν αναλυφθεί και μία βασική οπτική ε, γωνία η οποία κατά κάποιο τρόπο κατέστη το σημαντικότερο στοιχείο σε αυτή τη συζήτηση είναι ο ε, κίνδυνος, κυβερνοκίνδυνος με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Αυξάνεται φυσικά αυτός ο κίνδυνος στον κυβερνοχώρο και στην ε, τελευταία συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών ε, G7 ε, αποφασίσαμε ότι ήταν ένας από τους κυριότερους κινδύνους. Γι' αυτό ακριβώς οι εποπτικές αρχές υπησέρχονται στην όλη διαδικασία γιατί πρέπει να γίνονται επιθεωρήσεις που πρέπει να γίνεται κίνδυνος τεστ αντοχή σε τέτοιου είδου κινδύνου στο κυβερνοχώρο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καταστεί τρέχουσα πρακτική αυτό. Ε, βέβαια είναι περίπλοκο το ζήτημα και αυτό που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή είναι καταρχάς να υπάρχει μια εναρμονισμένη υποβολή εκθέσεων ε, ε, διαφόρων τέτοιων περιστατικών, κυβερνοπεριστατικών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ε, εποπτών κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας γιατί είναι σαφές ότι χρειάζεται συλλογική προσπάθεια ε, συλλογική προσπάθεια γίνεται ε, και σε παγκόσμιο επίπεδο, στο G7, στο G20 και στο BIS. Ελπίζω να σας κάλυψα. Είναι πάντως ένας τομέας που συνεχώς εξελίσσεται. Ευχαριστώ. Κύριε Λούκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τράκη. Ε, έχω τη χαρά σήμερα να μπορώ να θέσω δύο φορές ερωτήσεις σε εσάς. Θα ήθελα να επανάλθω στις ερωτήσεις ε, σας, ε, στην ερώτησή σας, στην προηγούμενη μου ερώτηση. Είπατε ότι, ότι τα νομισματικά μέτρα ε, σας συμμορφώνονται με την εντολή σας. Δεν κατάλαβα γιατί δεν βλέπετε να υπάρχει παραβίαση της απαγόρευσης της χρηματοδότησης κυβερνήσεων. Και υπάρχει παραβίαση της απαγόρευσης αυτής του άρθρου 123 της ε, συνθήκης εφόσον η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πιστωτής κυβερνήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, για αρκετά χρόνια. Γιατί λοιπόν δεν βλέπετε να υπάρχει τέτοια παραβίαση όταν ε, ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, παρέχει σημαντικές πιστώσεις στα κράτη-μέλη, αγοράζοντας ομόλογα, σε περίπτωση νέου δανεισμού των κρατών αυτών. Και μια ερώτηση σχετικά με την εντολή σας. Το PSPP ευνοεί τα κράτη-μέλη που έχουν υψηλά χρέη και υψηλά ελλείμματα. Το σύστημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ε, τα μεγαλύτερα δάνεια τα ε, έχει, ε, τα έχει παράσχει στις χώρες αυτές και αυτές οι χώρες έχουν ωφεληθεί περισσότερο. Γιατί αυτό θεωρείτε ότι συμμορφώνεται με την εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δύο σύντομες απαντήσεις. Καταρχάς, ε, δεν είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ακολουθούμε την ε, κλίδα κατανομής ε, κεφαλαίων. Και το είπα και πριν, το λέω και τώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει στις, στη δευτερογενή αγορά. Τρίτον, υπάρχει απόφαση του, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορείτε να εξετάσετε. Και τέταρτον, το PSPP αποτελεί αντικείμενο μιας προδικαστικής απόφασης ε, της, του δικαστηρίου που ζητήθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της ε, Γερμανίας. Όπως είχα ήδη τη δυνατότητα να διευκρινίσω, επειδή η ερώτησή σας αναφέρεται συγκεκριμένα στα θέματα αυτά που αποτελούν αντικείμενο απόφασης του ΔΕΚ, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω. Τέλος, όπως είχα τη δυνατότητα να ε, ε, εξετάσω και στο παρελθόν και κατά την τελευταία ακρόαση, θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων είναι νόμιμο, είναι σύνομο και εντός της εντολής μας. Ε, ο κύριος Λούκε, νομίζω ότι έχω χρόνο ακόμα. Πρέπει να προβλέψετε χρόνο όμως και για την απάντηση. Ναι. Ερώτηση σχετικά με το Target 2. Υπάρχει μηχανισμός εντός του συστήματος Target 2 που σημαίνει ότι οι ανισότητες εντός του, προγράμματος του συστήματος που δημιουργούνται μπορούν να ε, αντισταθμιστούν. Ε, ώστε να υπάρχει αντιστάθμιση ε, αναμέρα και επίσης ε, στις ε, αγορές αγαθών αλλά και αγορές κεφαλαίων των κρατών μελών. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός που οδηγεί σε αντιστάθμιση ή μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι ανισότητες, οι ανισορροπίες. δεν ήταν ο στόχος η επανεξισορρόπηση. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρο. και δεύτερον δεν αντικατοπτρίζουν ε, τα πλεονάσματα αυτά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Ιταλία έχει πολλά θέματα στα πλαίσια του Target 2. Η Γερμανία έχει πολλές διεκδικήσεις στο Target 2. Τότε κανονικά θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερο έλλειμμα σε σχέση με τη Γερμανία. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο. Το Target 2 είναι στην ουσία ρύθμιση όλων των μορφών πληρωμών και ε, υπάρχουν δυνατότητες εξαγοράς από πλευράς μας εκεί όπου υπάρχουν διαθέσιμα και όχι μόνο θεωρητικά εκεί όπου υπάρχουν πλεονάσματα σε σχέση με το συγκεντρωτικό όπως είπατε σύστημα δεν υπάρχει ένας μηχανισμός επανεξισορρόπησης τον οποίο εσείς εννοήσατε δεν έχει σχεδιαστεί ποτέ κάτι τέτοιο Καλό σας ευχαριστώ λέει ο κ. Γκουαλτιέρη κλείσαμε το νομισματικό διάλογο θα ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως το δεύτερο τμήμα της ανταλλαγής απόψεων με τον Μάριο Ντράγκη ως Προέδρου του ESRB, Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Όπως ξέρετε, το, σύστημα, το Συμβούλιο αυτό έχει δημοσιεύσει τους τελευταίους μήνες κάποια σημαντικά έγγραφα. Είχαμε ήδη μια ανταλλαγή απόψεων με την ιδιότητα, με τον κύριο Ντράγκη στα πλαίσια αυτής του της ιδιότητας τον μήνα Μάιο του 2017 και τώρα λοιπόν θα συνεχίσουμε τη συζήτηση σχετικά με τις μακροπροληπτικές πολιτικές, του συστημικούς κινδύνους και σχετικά με την πρόταση η οποία έχει γίνει πρόσφατα από πλευράς ε, του Συμβουλίου αυτού. Αρμοδιότητες λοιπόν ε, του ε, κυρίου Ντράγκη και του συστήματος. Έχει το λόγο ο κύριος Ντράγκη. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, κυρίες και κύριοι. Ε, με χαρά επανέρχομαι εδώ και θα σας απευθύνω το λόγο ως πρόεδρος του ESRB ε, για δεύτερη φορά φέτος. Από τότε που συναντηθήκαμε δημοσιεύσαμε την έκτη ετήσια έκθεσή μας που καλύπτει την περίοδο ανάμεσα στην 1η Απριλίου του 2016 και τις 31 Μαρτίου του 2017. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει ε, τις προοπτικές σχετικά με τον κίνδυνο, τις ε, μακροπροληπτικές αναλύσεις της ε, και συζητά τη συνεισφορά της στο πλαίσιο το μακροπροληπτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσης αναφέρεται και στη συνέχεια των προηγούμενων συστάσεων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο συναντήσεων που είχαμε σας ενημέρωσα για το τι περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση και γι' αυτό σήμερα θα συγκεντρώσω την προσοχή μου σε τέσσερα επιμέρους θέματα. Καταρχάς εξελίξεις στο πλαίσιο το μακροπροληπτικό ιδιαίτερα σε σχέση με αντικυκλικά μέτρα για το, μέσω του αποθέματος ασφαλείας, όπως επίσης τις συνέπειες του νέου IFRS 9, τη συνεισφορά του οργάνου μας στην διαμόρφωση της πολιτικής πέραν του τραπεζικού συστήματος και την παρέμβασή μας στην αγορά παραλόγων, να παραγόγων. να ξεκινήσω τώρα με τα αντικυκλικά μέτρα στα πλαίσια των ποσοστών αποθέματος ασφαλείας. Προσπαθούμε να καταστήσουμε εδώ τις τράπεζες πιο ανθεκτικές. Μπορούν να αυξήσουν στις καλές εποχές τα κεφάλαιά τους για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που μπορεί να αναφανούν αργότερα. Ε, αυτή η αντικυκλική αν θέλετε τρόπη αντιμετώπισης των προβλημάτων μέσω των αποθεμάτων ασφαλείας ε, έχουν αποδειχθεί ότι τα μέτρα, έχει αποδειχθεί ήδη ότι τα μέτρα ενίσχυσης των ισολογισμών των τραπεζών σε άσχημες εποχές πιέζει την οικονομία αυτό είναι κάτι το οποίο ε, χειροτερεύει την οικονομική κατάσταση και εξασθενεί ακόμα τους ε, ισολογισμούς των πιστοτικών ιδρυμάτων. Ενώ ε, το μέσο αυτό των αποθεμάτων ασφαλείας θα βοηθήσει την κατάσταση θα διευκολύνει τις τράπεζες να παρέχουν πίστοση στην πραγματική οικονομία. Είδαμε αρκετές μακροπροληπτικές αρχές να χρησιμοποιούν το μέσο αυτό. Η Σουηδία το έκανε από το 2015. Το 2017 η Τσεχία και η Σλοβακία έχουν αυξήσει ακόμα περισσότερο τα αποθέματα ασφαλείας και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι θα θέσει σε λειτουργία το περιθώριο αυτό το νέο το 2018. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης ο αριθμός των χωρών είναι έξι με την Νορβηγία και την Ισλανδία να ενισχύουν τις μακροπροληπτικές τους πολιτικές. Το 2014 το ESRB δημοσίευσε μια σύσταση σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τα κυκλικά αυτά μέσα. Οι συστάσεις αυτές υπογράμμισαν το πόσο σημαντικό είναι για τις αρχές που καθορίζουν ακριβώς το επίπεδο αυτών των αποθεμάτων ασφαλείας να έχουν μια σωστή πολιτική επικοινωνίας. Οι αποφάσεις για τα αντικυκλικά αυτά μέτρα είναι αρκετά νέες, αλλά η ε, ανακοίνωση και η ενημέρωση αυξάνει την προβλεψιμότητα των πολιτικών, των μακροπροληπτικών και βελτιώνει τις δυνατότητες εσωτερικής διαχείρισης. Σχετικά με τον τομέα των οικοδομών γενικά, ε, εμείς συζητήσαμε κάποιες συγκεκριμένες ε, πηγές ανησυχίας στον τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν συναντηθήκαμε τον προηγούμενο Νοέμβριο. Από τότε τα κράτη-μέλη έχουν βελτιώσει το πλαίσιο πολιτικής τους, ...την Αυστρία σαν παράδειγμα, έχουν πάρει συμπληρωματικά μέτρα, ιδιαίτερα για την κατοικία όπως τη Φιλανδία. Οι περισσότερες χώρες έχουν μέτρα τα οποία στοχεύουν τους κινδύνους στον τομέα της κατοικίας και πολλές χώρες χρησιμοποιούν επιπλέον μέσα στο policy mix το οποίο έχουν ε, μακροπροληπτικά μέτρα μαζί με τα μέτρα τα οποία αυξάνουν ε, την αντοχή των δανειστών. Εμείς στην παρούσα φάση κάνουμε μία ανάλυση του κινδύνου των αγορών ακινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εμπορικών αγορών. Έχουμε στοιχεία λοιπόν, κάτι το οποίο όμως δεν ξεκαθαρίζει ακόμα την μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των αγορών. Γι' αυτό όλες οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν τις συστάσεις μας. Ε, ε, το όργανο μας συνεχίζει να παρακολουθεί λοιπόν τους κινδύνους στο οικονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το βασικό φόρουμ για τις ευρωπαϊκές αρχές για τον συντονισμό των μέτρων και τη σύγκριση των εμπειριών. Να επανέλθω τώρα στα ευρήματα της έκθεσης του ESRB για την δημοσιονομική σταθερότητα και τις επιπτώσεις του IFRS 9 Ξέρετε ότι αυτά ξεκίνησαν η συζήτηση με ερωτήσεις τις οποίες εσείς μας θέσατε. Οι πιο σημαντικές αλλαγές του 9 είναι το πέρασμα από τις καταγεγραμμένες ζημίες στις αναμενόμενες απώλειες πίστοσης ε, για να καταμετρηθούν οι προβλέψεις απομείωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις προβλέψεις απομείωσης ενωρίτερα και να λάβουν υπόψη τους τα NPLs διασφαλίζοντας ότι ο τραπεζικός τομέας μπορεί να αποκατασταθεί πιο έγκαιρα και πιο συνολικά όταν αντιμετωπιστούν προβλήματα στο μέλλον. Μία ταχύτατη και στραμμένη προς τα εμπρός αναγνώριση των απολειών στον τομέα της πίστοσης αντιμετωπίζει άλλωστε και την κριτική που ασκείται για το λεγόμενο too little too late, πολύ λίγο και πολύ αργά. Αν μια αρνητική κατάσταση μπορεί να εντοπιστεί έγκαιρα, ο προκυκλικός χαρακτήρας μπορεί να μειωθεί και η, η απομείωση αν θέλετε των πιστοτικών δυνατοτήτων μπορεί να είναι μικρότερη. Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των ζημιών μπορεί να καθησυχάσει τις αγορές για την επάρκεια των κεφαλαίων, των πιστοτικών ιδρυμάτων, μπορεί να βελτιώσει την διαφάνεια και μπορεί να βελτιώσει και την αποτελεσματικότητα της τάξης που πρέπει να χαρακτηρίζει την αγορά. Γι' αυτό λοιπόν το IFRS 9 είναι ένα βασικό σημείο βελτίωσης σχετικά ιδιαίτερα με τα NPLs, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αντιδρούν με νέο τρόπο και να ενημερώνουν σωστότερα όταν έχουν στοιχεία για τέτοιου είδους προβλέψεις απομείωσης. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι προβλέψεις απομείωσης μπορεί να αυξηθούν σημαντικά και απότομα όταν χειροτερεύσουν οι οικονομικές συνθήκες, κάτι το οποίο θα προκαλέσει προκυκλικές επιπτώσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων το εύρος αν θέλετε ε, ε, των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες Δεύτερον, ο γεωργικός και τομιακός ε, τρόπος κατανομής των δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών και της ευαισθησίας που έχουν τελικά οι τράπεζες στον κύκλο δραστηριότητας. Και τέλος, η ορίμανση των δανείων αυτών. Η έκθεση ESRB αντιμετωπίζει κάποιες πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προκύκλικες επιπτώσεις. Το stress test μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μέτρηση των διακυμάνσεων των προβλέψεων απομείωσης έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν ποσοστά αποθέματος ασφαλείας στα capital buffers αν χρειαστούν. Αν οι τράπεζες μπορούν να αντέξουν ένα υποθετικά αρνητικό σενάριο θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν μέσω της έγκαιρης ε, αναγνώρισης των αναμενόμενων ζημιών στον τομέα της πίστοσης όπως αυτό απαιτεί άλλωστε το IFRS 9. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και στις δραστηριότητες μας στον μη τραπεζικό τομέα. Όταν συναντηθήκαμε για τελευταία φορά υπογράμμισε τη σημασία που έχει ε, ένα σωστό καθεστώς ανάκαμψης και εξυγίανσης των τραπεζών, όπως επίσης και των CCP, των κεντρικών αντισυμβαλωμένων, που παίζουν σημαντικό ρόλο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η SRB συνεισφέρει στον τομέα αυτό, εντοπίζοντας τους τομείς που μπορούν να λυθούν ή να αντιμετωπιστούν μέσω μακροπροληπτικών παρεμβάσεων. Σαν παράδειγμα η γνωμοθέτηση της ESRB για την πρόταση του Συμβουλίου υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές για τις τράπεζες και τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους. Όταν ένας κεντρικός αντισυμβαλόμενος έχει να αντιμετωπίσει δυσκολίες, όταν οι τράπεζες που τον συναποτελούν αν θέλετε έχουν προβλήματα. Ταυτόχρονα η δημιουργία ενός εναρμονισμένου πλαισίου ανάκαμψης για τον ασφαλιστικό τομέα είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Οι κανονικές διαδικασίες πτώχευσης μπορεί να μην είναι πάντα σύμβατες με την προστασία αυτών που έχουν ασφαλιστικά συμβόλαια και τους στόχους της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι πόροι διαθέσιμοι μπορεί να μην είναι επαρκείς για την διαχείριση της αποτυχίας ενός μεγάλου ενός μεγάλου ε, ασφαλιστικού οργανισμού στην Ολλανδία και την Γαλλία έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες πλαισίων αντιμετώπισης τέτοιου είδους πτωχεύσεων ε, ασφαλιστικών ε, ε, οργανισμών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Και η Ρουμανία έχει επίσης αναπτύξει ένα συνολικό πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης για τέτοιου είδους δυσκολίες μετά από τα προβλήματα που αντιμετώπισαν δύο μεγάλες ασφαλιστικές ρωμανικές εταιρείες το 2014 και το 2015. Τώρα να πω για την αγορά παραγόγων. Το ESRB επίσης συγκεντρώνει την προσοχή του στην ανάλυση και παρακολούθηση των αγορών παραγόγων στα πλαίσια των, των, των μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό θα πρέπει οι συναλλαγές να κατατίθενται και να εγγράφονται. Ε, το ΕΜΙΡ έχει δώσει στο ESRB πλήρη πρόσβαση ε, στις τράπεζες δεδομένων των καταγεγραμμένων ε, συναλλαγών των αγορών παραγόγων. Η συλλογή αυτού του είδους του μεγάλου επίπεδου αν θέλετε δεδομένων θα βελτιώσει τη διαφάνεια των αγορών παραγόγων για αυτούς οι οποίοι σχεδιάζουν την, τα πολιτικά μέτρα παρά τα τεχνικά προβλήματα τα οποία είναι παρόντα λόγω της μοναδικής φύσης αυτού του τύπου της πληροφορίας, τα δεδομένα αυτά ήδη αποδεικνύουν να είναι ε, χρήσιμα έτσι ώστε να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας των αγορών παραγόγων από συστημικής πλευράς. Για το λόγο αυτό το ESRB συγκεντρώνει την προσοχή του στην ανάπτυξη δεδομένων υποδομών και αναλυτικών μεθόδων έτσι ώστε να περάσουμε σε ένα πιο έγκαιρο και πιο λεπτομερές σύστημα παρακολούθησης των αγορών παραγόγων. Η προσπάθεια που κάνουμε στον τομέα αυτό είναι σε εξέλιξη και ελπίζω να επανέλθουμε σε αυτά όταν συναντηθούμε στο μέλλον. Αν υπάρχουν ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που αντιποκροθήκατε στο αίτημά μας. Είναι πολύ χρήσιμη η έκθεσή σας που αναφέρεται στη βελτίωση του πλαισίου. Είναι λοιπόν θέματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά. Brian Hayes, ο πρώτο ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Τράγκη, σας καλωσορίζω και πάλι ως Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Ε, δύο ερωτήσεις. Η μία είχε να κάνει με τα μακροπροληπτικά εργαλεία που έχουν τώρα πια οι τράπεζες ε, στη διάθεσή τους. Ε, χρειάζεται πότε-πότε επιπλέον κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας ε, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά και αναφερθήκατε ήδη σε κάποιες χώρες που έχουν ε, εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία. Ε, η Ιρλανδία, η χώρα μου και άλλες χώρες ε, πέρασαν ε, αρκετά εξαιρετικά περιστάσεις σύντομα. Αναφερθήκατε στις ελλείψεις στην συλλογή δεδομένων. Αναφερθήκατε στον τομέα ακινήτων στη χώρα μου και στις άλλες χώρες του προγράμματος. Πιστεύετε ότι ακόμη δεν έχουμε τα δεδομένα για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την ανάγκη για περαιτέρω αποθέματα ασφαλείας στις τράπεζες, ιδιαίτερα στις χώρες που πέρασαν τρομερούς κλειδονισμούς στον τομέα των τραπεζών τους. Και η δεύτερη μου ερώτηση ε, είναι ότι ξέρω... Θα ήθελα να ξέρω τι επιπτώσεις υπάρχουν στο μακροδημοσιονομικό περιβάλλον ε, και με την επιτυχία της ποσοτικής χαλάρωσης, ε, την οποία αναγνωρίζω. Μιλήσατε για κύκλο επενδύσεων, επενδυτικό κύκλο στην προηγούμενη σας ομιλία εδώ σήμερα. Και οι αποταμιεύσεις των οικοκυριών ε, μειώνονται εφόσον ε, γίνονται πιο προσβάσιμα, πιο φθηνά τα δάνεια. Φαίνεται ότι τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν αυτό. Βλέπουμε και στη χώρα μου να αποταμιεύουν περισσότερο, ενώ θα έπρεπε οι πολίτες να χρησιμοποιούν τα χρήματά τους για επενδύσεις. Ανησυχείτε ότι αυτά τα ποσοστά αποταμίευσης μπορούν να επηρεάσουν το βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον το οποίο όλοι θέλουμε να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την πρώτη σας ε, ερώτηση, πέρσι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ε, υιοθέτησε σύσταση για να καλυφθούν τα κενά στην ε, συλλογή δεδομένων και η σύσταση αυτή κάλυπτε ε, και τον τομέα των ε, κατοικιών και τον τομέα των εμπορικών ακινήτων. Ε, σημαντικά κενά στα δεδομένα συνεχίζουν να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, δεν έχουμε κοινά συμπεφωνημένους ορισμούς για κάποιους βασικούς δείκτες δείκτες όπως είναι τα χρέη σε σχέση με το εισόδημα και δεν έχουμε λοιπόν ε, συγκρίσιμα δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να θεσπίσει ένα πιο εναρμονισμένο πλαίσιο για την παρακολούθηση των εξελίξεων ε, στις αγορές ακινήτων ε, στην Ευρώπη και η σύσταση αυτή παρέχει μια σειρά εναρμονισμένων δικτών και οι εθνικές αρχές συστήνεται να παρακολουθούν τους κινδύνους που προκύπτουν από τον τομέα ακινήτων και να χρησιμοποιήσουν εναρμονισμένους δείκτες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνεται τακτική ε, συλλογή δεδομένων ε, για τους δείκτες αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουμε δύο ροές εργασίας για τη δουλειά αυτή. Η πρώτη είναι μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η άλλη είναι εντός της Eurostat. Η πείρα μας δείχνει ότι είναι δύσκολο να κλείσουμε τα κενά αυτά. Περιμένουμε, περιμένουμε να δούμε περισσότερο ενθουσιασμό από κάποιους από τους φορείς που μόλις ανέφερα, αλλά είναι σημαντικό, διότι η γενική κατάσταση, και αυτό είναι κάτι που έχω πει και σε άλλες περιστάσεις, θα πρέπει οι ρυθμίσεις, οι δημοσιονομικές και οι τραπεζικές ε, να ακολουθούν τις εξελίξεις και η πείρα της κρίσης μας έδειξε ότι όσο πιο πολύ διαβρύνεται η οικονομική πολιτική τόσο πιο σημαντικό είναι να έχουμε αυστηρή ρύθμιση των τραπεζών. Όσον αφορά τα χαμηλά επιτόκια, δεν έχω δεδομένα αναχώρα αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, αλλά η συνολική εικόνα είναι ότι είναι σταθερά. Δεν βλέπουμε αύξηση ούτε κυρίως μείωση. Τα χαμηλά επιτόκια λοιπόν, μέχρι τώρα τουλάχιστον, και συνολικά, διότι μπορεί βέβαια να κρύβονται εδώ οι πραγματικότητες σε διάφορες χώρες, ε, δεν βλέπουμε να ε, μας ανησυχεί η συμπεριφορά των αποταμιευτών. Η Περβάνς Περές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την ιδιότητά σας ως Προέδρου του ESRB αναφερθήκατε σε ζητήματα ε, τα οποία εξετάσατε εκ του σύνεγγυς στην ετήσια έκθεσή σας, όμως δεν αναφερθήκατε καθόλου στο θέμα του Brexit και στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην ε, οικονομική σταθερότητα και τον μακροοικονομικό κίνδυνο που θα μπορούσε να ε, συνεπάγεται. Δεν θέλω να μου πείτε τις συνθήκες του διαζυγίου. Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς ποιες θα είναι ακριβώς οι συνθήκες αυτές. Υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις που γίνονται ως προς τον αντίκτυπο που θα έχει το Brexit όχι μόνο στις χρηματοοικονομικές αγορές που είναι το μεγαλύτερο τμήμα όσον αφορά την δημιουργία ε, αξίας ε, ε, επί του οποίου θα έχει αντίκτυπο το Brexit. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι η δική σας ανάλυση του θέματος αυτού επειδή υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά την εξέλιξη των επιτοκίων, των επιτοκίων. Δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με το ίδιο ε, το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, το ESRB. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να ξανασκέφτεται τη λειτουργία του, της νέας αυτής δομής και στη διαβούλευση που είχε γίνει με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν αποφασιστούν περαιτέρω περαιτέρω μεταρρυθμίσεις του ESRB, ε, προέκυψε ένα κείμενο και το κείμενο αυτό εισάγει κάποιες μικρές αναπροσαρμογές όσον αφορά τη διοίκηση του ε, Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να διατηρηθεί το καλό επίπεδο λειτουργίας δεδομένης της εμπειρίας που έχει πλέον το Συμβούλιο ή θα θέλατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες ώστε η ε, διακυβέρνηση, ε, να, ε, η διακυβέρνηση του ESRB να εξελιχθεί περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καταρχάς να απαντήσω το πρώτο ερώτημα είναι σαφές ότι το Brexit ε, θα ε, δημιουργήσει μεγάλα ε, προβλήματα γιατί πρόκειται για μια χώρα στην οποία βρίσκονται τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αν όμως γίνει σωστή διαχείριση, έχω την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Το βασικό, η βασική ευθύνη μας είναι η σωστή διαχείριση αυτής της αλλαγής με το σωστό τρόπο, με μια σωστή ανακατανομή ευθυνών, χωρίς να τίθεται ένα ε, αμφιβόλο η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, της ενιαίας αγοράς. Βέβαια αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά αυτό ε, περιμένουν οι πολίτες ε, και των δύο πλευρών. Και αυτό μας ζητούν. Είναι πολύ νωρίς να πει κανείς κατά πόσο... Ε, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια πλατφόρμα ε, διαπραγμάτευσης. Ε. Όμως, για να σας δώσω ένα παράδειγμα ενός ζητήματος που αν ε, τύχει σωστής διαχείρισης... δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, η συνέχιση των συμβάσεων. οποιοδήποτε τομέα και αν διαλέξει κανείς στις χρηματοπιστωτικές αγορές, δεκάδες, εκατοντάδες ε, ε, συμβόλαια υπάρχουν, ε, υπάρχουν τα επιτόκια, υπάρχουν οι αντισυμβαλόμενοι, υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί τομείς, πάρα πολλοί τομείς, οποίους υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια συμβολέων, κάτι το οποίο ενδεχομένως να πρέπει να αλλάξει στην περίπτωση του του Brexit και βέβαια εξαρτάται από τους όρους ε, υπό τους οποίους ε, θα γίνει το Brexit. Αν μπορούν τώρα οι δύο πλευρές ε, να βρουν έναν τρόπο ώστε αυτή η διαδικασία αλλαγής να είναι ευκολότερη, Διαφορετικά η όλη διαδικασία προφανώς ε, θα έχει ως αποτέλεσμα κινδύνους ε, και ε, η χρηματοοικονομική αστάθεια μπορεί να είναι ένας από τους βασικούς κινδύνους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα έπρεπε και οι δύο πλευρές να κινηθούν προς μια διαχείριση που εξασφαλίζει μια ομαλή μετάβαση χωρίς να τίθεται ένα αμφιβόλο η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. Τώρα, εμείς σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι με τις, απο... με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής όσον αφορά την ε, μακροπροληπτική αναθεώρηση για το κομμάτι που αφορά το ESRB λαμβάνει υπόψη ε, την ε, ευρεία συμμετοχή, τον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνονται οι συζητήσεις, η εργασία του ESRB μόνο μία παρατήρηση έχουμε να κάνουμε επεκτείνοντας ε, την ιδιότητα μέλους στο ESSM και στο SRB ε, και με δικαίωμα ψήφου κιόλας ε, οι δύο πρόεδροι της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής και της Τεχνικής Επιτροπής δεν έχουν πια εκείνη δικαίωμα ψήφου. Και νομίζω ότι αυτό δεν ήταν ε, κάτι το επιθυμητό, δεδομένου ότι οι δύο ε, πρόεδροι είναι οι, μόνοι, μόνες, οι μόνες μη θεσμικές φωνές στο ESRB και έχουν συμμετάσχει σε πολύ σημαντικό βαθμό στις συζητήσεις μας από τότε που άρχισε να υπάρχει το ε, Συμβούλιο μας. Οπότε η βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο να δοθούν πίσω τα ε, δικαιώμα, το δικαίωμα ψήφου, να δοθεί πίσω το δικαίωμα ψήφου σε, αυτούς τους δύο, ε, ε, σε αυτές τις δύο ομάδες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριος Μαριάς. Η ερώτησή μου, κύριε Πρόεδρε, αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, όπως λέμε, τα NPLs. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή η οικονομική κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Λόγω του μνημονίου το 25% του ΑΕΠ έχει χαθεί. Το 40% του πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Η ανεργία αυτή τη στιγμή είναι στο 21%, αν και εσείς ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την υπολογίσατε την πραγματική ανεργία στο 31,3%. Επομένω, υπ' αυτού του όρου δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, διότι αυτό σημαίνει ότι τα distress funds, τα κοράκια όπως τα λέμε, θα αρπάξουν τα σπίτια των Ελλήνων αντί πινακίου φακής. Ήθελα λοιπόν την άποψή σας σε μια πρόταση. Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι περισσεύουν περί τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ από το τρίτο δανειακό πακέτο των 86 δις που πήρε η Ελλάδα. Δεν χρησιμοποιούνται. Από αυτά 19,5 δις περίπου θα πήγαιναν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Επομένω η πρότασή μας είναι πολύ απλή να δημιουργηθεί ένα δημόσιο ταμείο για κόκκινα δάνεια. Ένα ταμείο σωτηρίας των δανειοληπτών. Ύψους 4,5 δις ευρώ. Θα μπορούσε να αγοράσει κόκκινα στεγαστικά δάνεια ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και με αυτόν τον τρόπο τα κοράκια δεν θα αρπάξουν τα σπίτια των Ελλήνων, αλλά θα μπορούν μετά οι Έλληνες δανειολήπτες να πάνε σε αυτό το ταμείο και να αρχίσουν να αγοράζουν σιγά σιγά το δάνειό τους. Και επίσης κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσε στην Ελλάδα να εφαρμοστεί το κυπριακό μοντέλο. Δηλαδή να υπάρχει δικαίωμα προτίμησης των δανειοληπτών. Αντί μια τράπεζα να πουλήσει το δάνειό της στο 6, στο 10% σε ένα distress fund, θα μπορούσε αυτό να το αγοράσει ο ίδιος ο δανειολήπτης. Με αυτόν τον τρόπο και η τράπεζα θα έπαιρνε τα ίδια χρήματα που θα έπαιρνε ούτως ή άλλως και από το φαντ και ο δανειολήπτης θα μπορούσε ο ίδιος να μην χάσει το σπίτι του. Και θα μπορούσε φυσικά, αν δεν είχε και αυτά τα χρήματα, να ενισχυθεί από το Δημόσιο Ταμείο για τα κόκκινα δάνεια. Θέλω λοιπόν την άποψή σας στο ζήτημα αυτό, διότι σε λίγο ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και θα δημιουργηθούν τεράστια κοινωνικά προβλήματα στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς να σας πω ότι εμείς στο ESRB δεν συζητήσαμε ποτέ την κατάσταση των μη εξυπηρετουμένων δανείων στην Ελλάδα. Δεύτερον, θα έλεγα ότι τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που αποφασίζουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ταμεία, τα, τα χρήματα ε, που υπάρχουν στα ταμεία αυτά. Τρίτον, αν κάποιο αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τότε και άλλε χώρε έχουν τέτοιου είδου δάνεια. Οπότε, αν αυτό νομιμοποιεί την αξίωση, τότε και άλλε χώρε μπορεί να έχουν την αξίωση αυτή. Τέταρτον, πρέπει να κάνουμε τη διάκριση και νομίζω ότι η κυβέρνηση της Ελλάδα το κάνει αυτό. Ε, διάκριση μεταξύ διαφόρων κατηγοριών ε, υπάρχουν οι ε, φτωχοί, μετά Υπάρχουν ε, οι άνθρωποι που κατ' εξακολούθηση να πτωχεύουν και βεβαίω νομίζω ότι η διαχείριση, για τη διαχείριση των δανείων αυτών γίνεται τώρα αυτή η διάκριση. Δεν ξέρω τώρα ε, τι θα κάνουν τα κρατημέλη. Δεν ε, θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ούτε ε, το ESRB με ποιον τρόπο πρέπει να κινηθεί μια χώρα. Πάντω, αυτή τη στιγμή η διαχείριση που γίνεται από την κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει του πληστηριασμού με τι εγγυήσει και τα χέγγια για του φτωχού καλό είναι να συνεχίσουν, αλλά από εκεί πέρα τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να επιδοτήσουν τις τράπεζες ε, για να είναι λιγότερο επώδυνη κοινωνικά αυτή η κατάσταση. Ε, κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα θα έπαιρνε 86 δισεκατομμύρια ευρώ δάνειο. Όταν τελειώσει το πρόγραμμα θα περισσέψουν 25 δις. 19,5 δις θα πήγαιναν στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Επομένως το θέμα είναι 4,5 με 5 δις από αυτά να πάνε στη δημιουργία ενός Ταμείου Σωτηρίας των Δανειοληπτών, ενός Δημοσίου Ταμείου για κόκκινα δάνεια. Αυτό είναι θέμα που αφορά το Eurogroup και την Τρόικα. Αλλά βεβαίω αφορά και εσά και ω μέλο τη Τρόικα και ω ECB. Και θέλουμε να έχουμε μια άποψη πάνω σε, αυτό, σε αυτό το θέμα, διότι από εκεί ενδεχόμενα μπορεί να υπάρξει σωτηρία των δανειοληπτών. Δεν θέλω να συζητήσω τα πλεονεκτήματα αυτή τη πρωτοβουλία, ε, αλλά ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε η Τρόικα πλέον τα χρήματα αυτά, τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Τρεμόσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Ντράγη. Έχω μια ερώτηση σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, διότι κάποιες χώρες έχουν ακόμα υψηλά επίπεδα τέτοιων δανείων και αυτό αποτελεί πρόβλημα για την φερεγγιότητα πολλών ευρωπαϊκών τραπεζών. Από τη μία, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πολλά από αυτά τα δάνεια ε, προέρχονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από την άλλη, κάποιες από τις χώρες που επηρεάζονται περισσότερα από αυτά είναι ακριβώς οι χώρες με την ε, χειρότερη εφαρμογή της ε, τελευταίας οδηγίας πληρωμών. Δεν πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σωστά ε, αυτήν την ε, οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές, διότι κάποιες πολυεθνικές ε, δίνουν λογαριασμούς σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 200-300 μέρες πληρωμής αντί για 60. Πιστεύετε ή όχι ότι είναι σημαντικό, κάνω λάθος. Μήπως ε, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εξετάσει το θέμα αυτό. Θα συμφωνούσα απολύτως. Πολλές, πολλά από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων προέρχονται από την μεγάλη ύφεση και πολύ συχνά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πληρώνονταν όπως θα έπρεπε. Οι οφειλέτες δεν πληρώναν τα δάνεια τους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εσείς αναφερθήκατε στις πολυεθνικές, αλλά ούτε και οι κυβερνήσεις δεν πληρώναν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επί μήνες συχνά και χρόνια. Συμφωνώ απολύτως με την πρότασή σας. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές, αλλά είναι γεγονός ότι οφείλονται σε μη πληρωμή μεγάλων φορέων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ε, αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Thank you. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ τον κύριο Τράγκη. Η Κεντρική Τράπεζα ήδη από το 2016 λέει ότι οι μακροπιστωτικοί κίνδυνοι οφείλονται στους χαμηλούς ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης που με τη σειρά τους οφείλονται στην νομισματική πολιτική η οποία ακολουθήθηκε μέχρι τώρα. Τα προβλήματα λόγω ακριβώς του εύθραστου χαρακτήρα της οικονομίας έχουν χειροτερεύσει όπως ε, και κάποιες αποφάσεις που δημιουργούν προβλήματα ε, στις αγορές και φέρνω εδώ το παράδειγμα της Banco Popular της Ισπανίας και κάποιων Ιταλικών πιστοτικών ιδρυμάτων. Αυτοί οι τρόποι αντιμετώπισης ε, εξηγούν τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ε, εσείς ο ίδιος ε, κύριε Ντράγκη υπερασπιστήκατε άλλωστε και τις αλλαγές στον τομέα του εργασιακού δικαίου ε, στην Ισπανία αγνοώντας κύριε Ντράγκη τις κοινωνικές συνέπειες. Ακριβώς όμως βλέπουμε ότι οι χαμηλές αμοιβέ είναι αυτές που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση του οικογενειακού πλαισίου στην Ισπανία. Κοιτάξτε να απαντήσω στις δύο ερωτήσεις τις οποίες θέσατε. Καταρχάς, χαμηλές αμοιβέ και αν είναι κίνδυνος για τις τράπεζες. Αυτό ισχύει όλο και λιγότερο. Τα χαμηλά επιτόκια έχουν διαμορφώσει μια ισχυρή ανάκαμψη των οικονομικών συνθήκων και έτσι οποιασδήποτε συνέπειες είχαν στους ιστοσκελισμούς των τραπεζών τα χαμηλά επιτόκια αντισταθμίζονται από την μεγαλύτερη ρευστότητα και τους ισχυρούς πράγματι σήμερα ρυθμούς ανάπτυξης που βελτιώνει ποιοτικά τις πιστοτικές διαδικασίες, μειώνει τις ε, προβλέψεις ε, ζημιών και βελτιώνει την ανθεκτικότητα και τα ισχυρά χαρακτηριστικά του πιστοτικού συστήματος. Αυτή είναι η απάντησή μου στην πρώτη σας ερώτηση. Στη δεύτερη ερώτησή σας, να πω ότι οι πολιτικές μας κάνουν αντίθετα, το αντίθετο από αυτά τα οποία νομίζω ότι μας είπατε. Οι πολιτικές μας δεν πιέζουν προς τα κάτω τις αμοιβέ. Οι πολιτικές μας είναι ο καλύτερος τρόπος στήριξης των ονομαστικών μισθών να αρχίσουν να αυξάνονται πάλι. Οι πολιτικές μας είναι αυτές οι οποίες ακριβώς σωτήνουν ε, στην ε, μείωση ακριβώς αυτού του κενού στον τομέα της παραγωγής και που θα οδηγήσουν ε, στην βελτίωση του λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Για το αν τώρα οι δράσεις της ισπανικής κυβέρνησης, κοιτάξτε, δείτε ποια είναι η πραγματικότητα. Δείτε το πώς εξελίσσεται η απασχόληση στην Ισπανία. Δείτε τι θέσεις ε, εργασίας δημιουργούνται. Δείτε όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αγορά εργασίας στην Ισπανία. Είναι προφανές ότι δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε σε επίπεδο τομεακό, σε επίπεδο ταχύτητας και σε επίπεδο ποιότητας. Αλλά νομίζω ότι τα στοιχεία είναι γενικά ενθαρρυντικά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντράγκη. 30 δευτερόλεπτα, κύριε Μπεμέχο. Θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς θα πρέπει να αναθεωρήσετε τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήσατε και που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή στην απασχόληση στην Ισπανία. Να σας υπενθυμίσω ότι η αύξηση ε, της ε, απασχόλησης είναι χαμηλότατου επίπεδου, οι αμοιβέ είναι επίσης πάρα πολλές χαμηλές και αυτό εξηγεί και τα χαμηλότατα επίπεδα παραγωγικότητας στην Ισπανία που δεν επιτρέπουν και δεν δικαιολογούν την Ισπανική κυβέρνηση να παίρνει τέτοια μέτρα. Είναι αλήθεια ότι η ονομαστική μισθή ε, αλλάζουν με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Γιατί η παραγωγικότητα είναι χαμηλή, αυτό ισχύει για την Ισπανία αλλά και για άλλες ε, χώρες. Εδώ η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να κάνει τα πάντα μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση με χαμηλά επιτόκια, υψηλότερη κατανάλωση και υψηλότερες επενδύσεις. Αυτό επηρεάζει τις θέσεις απασχόλησης αλλά όχι την ποιότητα της απασχόλησης. Δεν είναι όμως αυτή η δουλειά της νομισματικής πολιτικής. Όσο όμως αναπτύσσονται, ε, ε, όσο αναπτύσσεται η οικονομία θα βελτιώνονται και οι αμοιβέ. Και επίσης ε, μπορούμε λίγο να επηρεάσουμε την παραγωγικότητα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε και βοηθάμε να γίνουν, αλλά υπάρχουν και πράγματα που δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες των κεντρικών τραπεζών. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κόμπερν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Ντράγκη. Είχατε πει παλαιότερα ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες η επιστροφή στον προστατευτισμό θα δημιουργούσε κινδύνους στην παγκόσμια οικονομία. Πράγματι, ο προστατευτισμός δημιουργεί προβλήματα στη σταθερότητα του πιστοτικού συστήματος. Δεν ξέρω, μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε και κάποιες μελέτες κατά περίπτωση. Έχετε υπολογίσει σαν παράδειγμα τι συνέπειες θα έχει στο ισπανικό χρέος η αποχώρηση της Καταλωνίας. Η Καταλωνία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του ισπανικού ΑΕΠ, θυμίζω. Και δεύτερον, ποιες θα είναι οι συνέπειες ε, του Brexit στο εύθραυστο ε, τραπεζικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα Γαλλία και Ιταλία. Αυτές οι χώρες ε, θα χτυπηθούν άσχημα από τη μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Δεν μπορούμε με μέτρα προστατευτικά να καλύψουμε την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν μπορούμε να καταστήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της ευρωπαϊκής οικονομίας πιο ακριβό και πιο ακριβή την δυνατότητα χρήσης των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών. Το 85% έτσι και αλλιώς των κεφαλαίων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνούν από το Λονδίνο, οπότε οι οικονομίες κλίμακας θα πρέπει να γίνουν στο Λονδίνο ε, η επενδυτική τράπεζα του η επενδυτική τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Λονδίνο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να παίρνετε μέτρα που να, να δημιουργούν προβλήματα στην σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει νομίζω το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου όλα αυτά τα θέματα να ανταλάβει υπόψη του σοβαρά. Θα συμφωνήσω μαζί σας λέγοντας ότι το Brexit είναι ε, ένα σημαντικό υπαρξιακό αν θέλετε συμβάν του οποίου οι συνέπειες θα πρέπει να συζητηθούν και να αναλυθούν προσεκτικά. Γιατί δεν το έχουμε κάνει ακόμα αυτό ή τουλάχιστον το ESRB δεν το έχει κάνει γιατί δεν έχουμε μια ακριβή άποψη, έστω και ανακριβή αν θέλετε, του ποια θα είναι η πλατφόρμα διαπραγμάτευσης. Γνωρίζουμε ότι το μέγεθος των αγορών είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Σε όλους τους τομείς των χρηματαγορών, είτε στις τράπεζες σαν παράδειγμα, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, ποσοτικά στοιχεία τα οποία είναι υψηλού επίπεδου και θα πρέπει να τύχουν της προσοχής μας ανάλογα με τον τρόπο που θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις. Όπως είπα, η μετάβαση αυτή μπορεί να γίνει αντικείμενο διαχείρισης με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές πλευρές. Αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει να μην θέσει σε κίνδυνο ε, την, τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της εσωτερικής αγοράς. Βέβαια τα λόγια εδώ είναι εύκολα και ε, έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι μέρος ε, της διαπραγματευτικής ομάδας. Πάντως η δουλειά που έχουμε μπροστά μας όλοι είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Θα δούμε λοιπόν πώς οι δύο πλευρές προχωρούν στις διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια καλύτερη αντίληψη, θα κάνουμε την πρώτη συζήτηση και το ESRB είναι ένα ιδανικό φόρουμ για συζήτηση. Δεν περιορίζεται στην Ευρωζώνη, δεν περιορίζεται σε κάποιες τράπεζες ή ε, νομίζω ότι ε, και υπάρχουν και ανεξάρτητες φωνές αυτοί που ηγούνται των δύο επιτροπών του ESRB. Νομίζω ότι η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα είναι θα έλεγα ενδιαφέρουσα. Μου φαίνεται ότι ο κύριος Μπαρνιέ και ο κύριος ε, με, με, ε, ε, Φερχόφστατ ουσιαστικά είναι δύο αυτοκίνητα που κοιτάνε ο ένας τον άλλον και βλέπουν ποιος θα, φο, ποιο θα το ένα το άλλο και ποιο θα φοβεί το άλλο. θέλετε να τιμωρήσετε τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, πολύ επικίνδυνο και για την Ισπανία και για την ε, οικονομία της Ευρωζώνης και ίσως θα έπρεπε να πείτε στον κύριο Φερχόφστατ και στον κύριο Μπαρνιέ να, βρείτε, να βρούνε μια λύση. Όπως ξέρετε, και εγώ συμμετέχω στην ε, ομάδα αυτή με τον κύριο Φερχόφστατ, ε, δεν έχουμε καμία τιμωρητική διάθεση. Εμείς θέλουμε μία δίκαιη ε, συμφωνία που θα είναι αποφελής για τους. Ελπίζω να τους μιλήσετε πάντως. Ελπίζω να τους μιλήσετε, λέει ο κύριος Κόμπουν. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Μάρκο Τζάνι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Τράγκη. Ξέρετε ότι το θέμα των κρατικών ομολόγων που επιβαρύνουν κάποια πιστοτικά ιδρύματα είναι αντικείμενο συζήτησης. Έχουν γίνει αρκετές ανεπίσημες συζητήσεις, έχουν γίνει κάποιες προτάσεις γύρω από τις οποίες ε, η συζήτηση προχωράει και σε σχέση με την ε, δυνατότητα εγγύησης των καταθέσεων που υπάρχει μια αναζήτηση ε, της, του σωστού τρόπου μείωσης του κινδύνου για τους καταθέτες. Γνωρίζετε ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δημοσιεύσει πρόσφατα τις κατευθυντήριες γραμμές για τα stress test του 2018 και η αξιολόγηση των κρατικών ομολόγων και του κινδύνου που μπορεί να αποτελούν στις τράπεζες θα ληφθεί υπόψη. Το ερώτημά μου λοιπόν αφορά τον δυνητικό κίνδυνο για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα μπορούσε να προκληθεί από το θέμα που προανέφερα στα πιστωτικά ιδρύματα. Από τη μία θα μπορούσε να υπάρξει μια προληπτική αν θέλετε διάθεση συμπληρωματικών κεφαλαίων για τις τράπεζες οι οποίες κατέχουν τέτοιου είδους κρατικά ομόλογα διαφορετικού επίπεδου και διαφορετικού κινδύνου και από την άλλη να υπάρξει ένα ανώτατο όριο στην αγορά τέτοιου είδους ομολόγων από πλευράς των τραπεζών. Είναι κίνδυνοι λοιπόν αυτοί ε, που μπορεί να δημιουργηθούν για τις τράπεζες. Ε, καταρχάς το θέμα της ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι εν κινδύνο. Ξέρετε ότι τα κρατικά ομόλογα είναι ένα collateral πολύ σημαντικό και σε σχέση με τα ρέπος και μπορεί να επιρεώσει την ρευστότητα και τελειώνω εδώ πρόεδρε λέγοντας ότι πρέπει να παρατηρήσουμε και την πιθανή πίεση που μπορεί να ασκηθεί στα κρατικά ομόλογα ορισμένων χωρών και σε ορισμένες χώρες των οποίων τα πιστοτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Οπότε θα πρέπει οι τράπεζες ή να ξεφορτωθούν σε εισαγωγικά ε, τέτοιους κρατικούς τίτλους ή διακόπτει ο Η θέση, η θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το θέμα αυτό είναι κατόπιν ε, μελετών και από το ESRB και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επί του θέματος αυτού είναι ε, καταρχάς αν υπάρχει ένας κίνδυνος θέλουμε να μειώσουμε τη σχέση μεταξύ του δημοσίου χρέους ε, και ε, των προβλημάτων των, ε, τραπεζών, των ισολογισμών των τραπεζών. Το πώς θα το κάνουμε αυτό βέβαια είναι κάτι διαφορετικό. Ε, οποιασδήποτε συμφωνίες, οποιοδήποτε συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξουμε ε, ένα είναι βέβαιο, δεν θέλουμε να έχουν ε, συγκριτικό μειονέκτημα οι δικές μας τράπεζες σε σχέση με τις τράπεζες όλου του υπολείπου κόσμου. Γι' αυτό λαμβάνουν χώρα μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις στην Επιτροπή Βασιλεία, Βασιλείας και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει συνένεση για ε, ε παγκόσμια συμφωνία επί του θέματος αυτού. Χώρες δηλαδή άλλες χώρες δεν συμφωνούν με ε, σταθμίσεις ή περιορισμούς. Οποιαδήποτε τώρα συμφωνία στην οποία ενδεχομένως να καταλήξουν οι Ευρωπαίοι, αν υπάρξει ε, τέτοια συμφωνία, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τρεις λοιπόν ε, προϋποθέσεις. Να μην υπάρχουν ε, σκληροί περιορισμοί, πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη συμφωνία. Αν οι Ευρωπαίοι πρέπει να κινηθούν μόνοι τους, η συμφωνία πρέπει να εφαρμοστεί ε, σωστά και όπως πρέπει. Κάτι ακόμη θα ήθελα να ρωτήσω. Εσείς είπατε σωστά ότι οι ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να βρουν μια κάποια συμφωνία για τη μη δημιουργία στρεβλώσεων στην αγορά αυτή. Πώς ε, είπε και ο Μπενουά το 16 ε, η κατάσταση των κρατικών ομολόγων στην, ε, στα, στις, στις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό της Ευρωζώνης γιατί φυσικά σε ε, μια χώρα η οποία ελέγχει ξεκάθαρα το νόμισμά της τέτοιου είδους τίτλοι δεν αποτελούν σημαντικό πρόβλημα. Συμφωνώ απολύτω. όμως αυτή η συμφωνία δεν ε, έχει υπάρξει ακόμη και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί αν η Ευρώπη αποφασίσει να κινηθεί ε, με το δικό της τρόπο, τότε θα έπρεπε να γνωρίζει ότι τέτοιου είδους μέτρα θα μπορούσαν ε, να ε, δημιουργήσουν ένα συγκριτικό μειονέκτημα στις ευρωπαϊκές τράπεζες σε σχέση με τις ε, τράπεζες του υπολοιπού κόσμου. Γι' αυτό ακριβώς μια παγκόσμια συμφωνία θα ήταν προτιμητέα. Αυτή είναι και η άποψη του Κοινοβουλίου, λέει ο Πρόεδρος, στο πλαίσιο της Βασιλείας. Ο κύριος Κύρτσος. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και τι γίνεται με το συστημικό κίνδυνο που αφορά τον τομέα των ακινήτων. Μιλούμε για έναν αναχώρα κίνδυνο, έναν κίνδυνο σε επίπεδο χώρας ή μιλάμε για ένα πολύ τοπικό ε, συγκεκριμένο κίνδυνο. Και το άλλο ερώτημα που είναι μάλλον πολιτικού χαρακτήρα αλλά θεωρώ ότι είναι καθήκον μου να σας το θέσω έχετε μία ανυφάλια προσέγγιση προς το συστημικό κίνδυνο, αλλά δεν έχετε το φόβο ότι θα είστε λίγο μόνος στο μέλλον, γιατί υπάρχει μεγάλη πολιτική αβεβαιότητα. Ε, το Brexit, για παράδειγμα, δεν ξέρει κανείς πώς θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις. Στη Γερμανία και στην Αυστρία ε, οι συνάδελφοι δεν είναι εδώ γιατί φαντάζομαι ότι προσπαθούν να δουν ε, ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα τους. Ε, έχουμε λοιπόν αυτή την, αντίφα... την ε, διαφωνία μεταξύ Μαδρίτης και Καταλωνίας. Ε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει, από παράδειγμα, στην Ιταλία σε επόμενες εκλογές. Υπάρχει λοιπόν μια πολιτική αστάθεια. Αυτή η πολιτική αστάθεια θα μπορούσε να δημιουργήσει οικονομικούς και συστημικούς κινδύνους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία οικονομικής εξέλιξης από την πολιτική κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στο δεύτερο σας ερώτημα πρώτα. Η δική μας εμπειρία των τελευταίων δύο ετών είναι η αντίστροφη. Ε, θα θυμάστε ότι προβλέπονταν τρομερές καταστροφές ε, μετά το Brexit, ε, μετά τις εκλογές σε σημαντική χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απειλητική κατάσταση προβλεπόταν όσον αφορά τις εκλογές σε μία συγκεκριμένη χώρα και ούτω καθεξής. Ε, η εμπειρία μας όμως μας έδειξε ότι η ανάκαμψή μας είναι ισχυρή, είναι ανθεκτική και μπορεί να αντέξει ε, κάποιον από αυτό το κίνδυνο. Βέβαια, ε, δεν έχουμε κρυστάλλινη σφαίρα για να προβλέψουμε το μέλλον και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει και κατά πόσο υπάρχει περίπτωση να ε, ε, προκληθούν ε, κίνδυνοι που θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην ανάκαμψη, αλλά μέχρι τώρα είναι θετικά τα πράγματα. Κάτι ακόμη με ρωτήσατε. Η έκθεσή μας αξιολογεί ο κυρίως τα κίνητα κατοικίας και θεωρεί ότι οι τιμές είναι αρκετά υψηλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και υπήρξαν και οκτώ αναχώρα ειδικέ προειδοποιήσεις και εντοπίζουν μεσοπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα προβλήματα στον τομέα αυτό των ακινήτων κατοικίας. Και αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα των νοικοκυριών να πληρώσουν τα χρέα τους και κάποια, τα χρέα τους και κάποια άλλα από την εξέλιξη της δυναμικής των τιμών των ακινήτων κατοικιών. Οι χώρες ε, σε γενικές γραμμές ανταποκρίθηκαν με μέτρα στη Δανία και στη Φιλανδία για παράδειγμα, άλλαξαν τη στάθμιση κινδύνου, στη Σουηδία επίσης ε, ε, υπήρξαν κάποια κίνητρα απόσβεση των δανείων, ε, αλλά σε γενικέ γραμμέ είναι αρκετά υψηλέ οι τιμέ. Ε, τελευταία ερώτηση, ο κύριο Μορκάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για την παρουσία σα εδώ κύριε Ντράγκη. Καταρχά τα λεγόμενα SBBS, εγγυημένα ευρωπαϊκά ομόλογα, τα οποία είναι υπομελέτη από την Επιτροπή σας. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής πρέπει να κυκλοφορήσουν ε, πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα και υποτίθεται ότι θα ακολουθήσει μια νομοθετική πρόταση από πλευρά πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να μάθω πώς η Επιτροπή αυτή μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι θα είναι ασφαλής η τίτλη αυτή. Θα είναι τριπλό αλφα δηλαδή και ταυτόχρονα πώς μπορεί να διασφαλίσει ότι η αγορά των τίτλων αυτών θα έχει επαρκείς διαστάσεις και επαρκή ρευστότητα. Πιστεύετε ότι η δημιουργία αυτού του τύπου των ομολόγων <clears throat> μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα κρατικά ομόλογα και ε, τη σταθερότητα γενικότερα στις χώρες της Ευρωζώνης. <clears throat> Υπογραμμίσετε επίσης τη σημασία που έχει η μείωση των NPLs. Το θέμα είναι πόσο μπορούμε να το πετύχουμε αυτό αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσουμε μέτρα τα οποία θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις συνολικά στην αγορά των NPLs ή συμφωνείτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θέλει να υπάρξει ένας συνδυασμός μέτρων και νομοθετικών και περιορισμού των νέων δανείων. Εδώ ήμουν λίγο συνοπτικός, συγγνώμη για την ταχύτητα. Θα απαντήσω στα αγγλικά. Θα συμφωνήσω με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το είχα πει και παλαιότερα εδώ και λίγο καιρό. Είχα πει ότι αυτό το οποίο απαιτείται είναι μια κοινή προσπάθεια από πλευράς όλων των εμπλεκομένων των εποπτικών αρχών, των πιστοτικών ηρημάτων και των κυβερνήσεων που θα πρέπει να δώσουν την δυνατότητα δημιουργίας του επαρκούς νομοθετικού πλαισίου έτσι ώστε τα NPLs να μπορέσουν να τα μειώσουμε. Συνεπώς λοιπόν όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, των μη εξυπηρετούμενων δανείων, έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα και να μην δημιουργηθούν αποστεθεροποιητικές επιπτώσεις όπως αυτές τις οποίες είπατε ότι φοβάστε. Οπότε θα συμφωνήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Για το άλλο σας ερώτημα, να ξεκινήσω λέγοντας ότι απαιτείται ε, μια, ασφαλ, ένας ασφαλής τίτλος. Ε, είναι κάτι το οποίο χρειάζονται οι ίδιες οι αγορές. Η αναζήτηση ενός τέτοιου τύπου τίτλου είναι δικαιολογημένη. Τώρα, αν αυτό το συγκεκριμένο μέσο, το SBBS, ε, ανταποκρίνεται σε αυτή την αναζήτηση, αυτό θα το συζητήσουμε και θα δούμε ακριβώς τι θα κάνουμε με τη μελέτη η οποία θα κυκλοφορήσει, αν θα κυκλοφορήσει, με ποια μορφή κτλ. Και θα εξετάσουμε ποιο είναι το επόμενο βήμα μας. Πάντως, νομίζω ότι οι εργασίες αυτές θα συνεχιστούν, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, απαιτείται η ύπαρξη ενός ασφαλούς τίτλου μιας μορφής τίτλου δηλαδή που να παρουσιάζει τα ηχέγγυα ασφάλεια που επιθυμούμε. Τώρα θα πρέπει να αλλάξουμε κάτι το οποίο υπάρχει, εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια μακρά, αλλά νομίζω πολύ χρήσιμη συζήτηση. Πρόεδρε Ντράγκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε εδώ να συνομιλήσετε με τα μέλη της Επιτροπής μας για μια σειρά ζωτικών θεμάτων ε, για ε, τις δημοσιονομικές προοπτικές μας. Σας ευχαριστώ πολύ.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

Okay. Α, περνάμε στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Uh, μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ιδίων Πόρων. Έχουμε την παρουσίαση της πρότασης ψηφίσματος για τη γνωμοδότησή μας. Ο Λουίτζι Μόργανο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τους συναδέλφους που είναι εδώ και ιδιαίτερα τους σκιώδεις εισηγητές. Θα έχετε όλοι διαβάσει το σχέδιο γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Και γι' αυτό θα επανέλθω στα βασικά σημεία. Το θέμα της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και όχι μόνο λόγω του Brexit. Τίθεται το θέμα υπευθυνοποίησης των ευρωπαϊκών οργάνων στην ουσία χρησιμοποιώντας ε, αυτά τα οποία έλεγαν στο Boston Tea Party καμία αντιπροσώπευση, καμία φορολογία. Στόχος δεν είναι η αύξηση της φορολογίας εις βάρος των πολιτών, αντίθετα όμως να απελευθερώσουμε πόρους οι οποίοι μπορεί να γίνουν αντικείμενο διαχείρισης με πιο δημοκρατικό τρόπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μειώνοντας τον προϋπολογισμό των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης ή τουλάχιστον να μην αυξηθεί αυτός. Προτείνουμε λοιπόν κάποιους ίδιους πόρους για την Ευρωζώνη και κάποιους πόρους πιο συγκεκριμένους ε, που καλύπτουν τις δραστηριότητες της Ένωσης. Σαν παράδειγμα σε επίπεδο Ευρωζώνης να υπάρξει μια μορφή φορολογίας για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και μια φορολογία για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αγορές κεφαλαίων. Βασικός στόχος είναι να διευκρινίσουμε με καλύτερο τρόπο τη σχέση ανάμεσα σε χρηματοδότηση και δαπάνη στον Ευρωπαίο προϋπολογισμό και να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε και νέους πόρους για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Δεύτερον, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, να μάλλον ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν από την Ευρώπη ως κοινότητα και όχι σαν σύνολο κρατών μελών την καταπολέμηση της ανεργίας, την προώθηση των επενδύσεων, την εγγύηση των εξωτερικών συνόρων και αυτά τα κοινά ευρωπαϊκά αγαθά δεν μπορούν να, ευρωπαϊθούν, να ολοκληρωθούν με μέσα τα οποία δεν ελέγχονται δημοκρατικά από τις συνομοθέτες. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι πρέπει να διευκρινίσουμε καλύτερα πώς τα δημόσια αυτά αγαθά, τα οποία εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Επιτροπή μας, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με τους ίδιους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Τέλος, όπως και σε εθνικό επίπεδο συχνά, ε, υπάρχει μια πτυτικότητα θα έλεγα σε σχέση με τον οικονομικό κύκλο. Το θέμα δεν είναι ε, να χειροτερεύσουμε την κατάσταση στα κράτη-μέλη που έτσι και αλλιώ υφίστανται κάποιους περιορισμούς σε σχέση με το χρέος και το έλλειμμα. Πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να αποφύγουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποια ιδιοσυγκρατικά στοιχεία τα οποία λειτουργούν αρνητικά σε εθνικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάλετιτς από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Λουίτζι Μοργάνο, για το, το σχέδιο γνωμοδότησής του. Νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε μια πολύ σημαντική πρόκληση. Με το Brexit ε, θα μειωθεί ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωσης και θα σκεφτούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις νέες προκλήσεις. Μάλιστα ούτε καν στις καινούριε μόνο, αλλά μιλάμε για την άμυνα, ε, την ε, μετανάστευση, πώς θα ενισχύσουμε την Ευρωζώνη, πώς θα ενισχύσουμε την ενιαία αγορά και ένα σωρό άλλα θέματα. Ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσουμε και τις υπάρχουσες πολιτικές. Για παράδειγμα, η πολιτική συνοχή θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και όχι να αποδυναμωθεί, διότι χρειαζόμαστε πραγματική σύγκληση των χωρών που βρίσκονται πιο πίσω, εάν θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή νομισματική Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Οι αποφάσεις λοιπόν σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι εύκολες. και με το Brexit και το γεγονός ότι θα συρρυκνωθεί ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν θέλουμε να ενισχύσουμε τον προϋπολογισμό, θα πρέπει είτε να εισάγουμε νέους πόρους είτε να αυξήσουμε τις ε, ισχύουσες συνεισφορές. Εξετάζοντας λοιπόν τώρα την πρόταση της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου για τους ίδιους πόρους, η ομάδα αυτή προσπαθεί να έχουμε ένα πιο δίκαιο, διαφανές και αυτόνομο σύστημα, κάτι που θα θέλαμε και εμείς να δούμε, και προτείνει μείωση του ε, ποσοστού του ΑΕΠ να είναι πιο αυτόνομος ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, προτείνει επίσης κατάργηση του διορθωτικού μηχανισμού, απλούστευση δηλαδή. Επίσης, μεταβίβαση ε, ενός ε, ποσοστού του ΦΠΑ και κάτι που συζητήσαμε μόλις τώρα με τον κύριο Ντράγκη. να στηρίξουμε ή όχι τμήμα του κέρδους Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μπαίνει στον προϋπολογισμό. Επίσης, φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικές αποφάσεις που θα πρέπει να λάβουμε και θα πρέπει να αναλύσουμε την σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα όλων των συστάσεων αυτών και να σκεφτούμε ποια θα πρέπει τελικά να είναι η οριστική πρόταση την οποία θα ε, μεταφέρουμε στους πολίτες μας, διότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα στις μέρες μας, ε, διότι έχουμε ακόμη ανάπτυξη αργή, όμως οι προβλέψεις ε, φαίνονται θετικές, έχουμε όμως ακόμη χαμηλή παραγωγικότητα, γι' αυτό δεν έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση μισθών, γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και την αντίδραση του κοινού στις τροποποιήσεις ε, του συστήματος ιδίων πόρων που ε, σημαίνει είτε εισαγωγή νέων φόρων είτε αύξηση της εθνικής συνεισφοράς. Ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε τι ωφέλη θα έχει και για τους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Λίδη Βίρνικ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Μιλώ εκ μέρου ε, του Ενρίκα Καλκχάφτουμ, Κύριε Σιγητά, κύριοι σκιώδη εισηγητέ, πιστεύω ότι ο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεωρείται ένα μέσο κοινή πολιτική για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων, όπω επίση και για την, ε, το συντονισμό ε, των προσπαθειών ε, για την, αύξηση, για την ανάπτυξη και για την αύξηση της απασχόλησης ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έναν επενδυτικό κύριο προπολογισμό, η ευελιξία και ε, η δυνατότητα παρέμβασης ε, βραχυπρόθεσμης είναι, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ο προπολογισμός είναι πολύ μικρός ε, για πραγματική και ε, αντικυκλική σταθεροποίηση ως πραγματικός υποστηρικτής ε, ε, της αναθεώρησης αυτής θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του συστήματος των ιδίων πόρων με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα βασικά μέσα που προτείνει ο εισηγητής μπορεί να βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς αν μειώσουν την, τον ε, ε, πολλαπλασιασμό των φόρων με συντονισμένο τρόπο και θα υπάρξει μια σχέση έτσι μεταξύ ε, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και των πολιτικών της Ένωσης. Η αναθεώρηση του ΦΠΑ είναι πάρα πολύ σημαντική, χρειάζεται μεγαλύτερη εναρμόνιση προκειμένου να προωθήσουμε δικαιότερη φορολόγηση και αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, ε, επιπλέον βέβαια της χρηματοδότησης του ενωσιακού προπολογισμού. Θα υποβάλω τροπολογίες για να μπορέσω να ε, τονίσω για παράδειγμα ε, το πόσο αναγκαίο είναι να υπάρχει ένα πραγματικό νομισματικό ταμείο που να βασίζεται σε ενωσιακό δίκαιο και με πολύ χαρά θα συζητήσω το θέμα αυτό και με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εξ ονόματος του Μιγγέλ Βιέχας που είναι σκιώδης εισηγητής ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα εδώ. Εμείς θεωρούμε πάρα πολύ θετική την έβρεση νέων τρόπων φορολογίας για τις συναλλαγές σε επίπεδο χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Πάντως θεωρούμε ότι η συζήτηση αυτή θα πρέπει να, να ενταχθεί στα πλαίσια της συζήτησης για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό έτσι ώστε να υπάρχουν συνεισφορές προς τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό από τις διάφορες χώρες με βάση το εθνικό σύστημα γιατί αλλιώς η χρησιμοποίηση φόρων όπως το ΦΠΑ είναι κάτι το οποίο επιτείνει τις ανισότητες ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Απαιτείται επίσης η αναδιάρθρωση, η μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης σε σχέση με την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Υπουργείου Οικονομικών και να μην γίνονται ε, ε, προσπάθειες επιρροής των κρατών μελών ή των υποψηφίων χωρών έτσι ώστε να λαμβάνουν νεοφιλελεύθερα μέτρα με ε, αλόγιστες κοινωνικές συνέπειες και δεν θα πρέπει επίσης να υφίστανται οι χώρες αυτές εκβιασμούς για τη διάλυση του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον ε, εισηγητή για τη δουλειά του πάνω στη γνωμοδότηση αυτή που ακολουθεί μια κατεύθυνση που μπορεί να στηρίξουν και οι πράσινοι. Βλέπουμε δηλαδή ε, με επικριτικό μάτι την αντικατάσταση του, του τμήματος ε, ναι, που βασίζεται στο ΑΕΠ από ίδιους πόρους. Βέβαια μπορούμε να σκεφτούμε και έσοδα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ε, θα τα εξετάσουμε όλα αυτά. Θα προσθέσουμε και μία τροπολογία που θα εξετάζει τι θα γίνεται με τα πρόστιμα που θα πληρώνονται με βάση αποφάσεις ε, του ΔΕΚ, ε, το οποίο μπορεί και αυτό να αποτελέσει ίδιο πόρο. Γενική υποστήριξη λοιπόν ε, για τη γνωμοδότηση του ε, συντάκτη. Σίγουρα η πράσινη είναι υπέρ του να είναι πιο σαφές το σύστημα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μία ερώτηση έχουμε μόνο στην παράγραφο 4 όπου ο εισηγητής ε, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδει χρεόγραφα μηδενικού κινδύνου προκειμένου να αντισταθμίζει την αστάθεια των εσόδων από ιδίου πόρου. Αναρωτιόμαστε, αυτό είναι δυνατόν χωρί τροποποίηση τη ε, συνθήκης, διότι σύμφωνα με τη συνθήκη δεν επιτρέπεται να χρεωθεί η Ένωση. Μια ερώτηση γι' αυτό κατά τα άλλα στηρίζουμε τον εισηγητή και θα ενισχύσουμε κάποια τμήματα της ε, γνωμοδότησης. Γενικά όμως τη στηρίζουμε. Ε, όπως γνωρίζετε το EFSM μπορεί να εκδώσει χρεόγραφα. Αυτό βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά είναι κάπως πιο πολύπλοκο το θέμα. Ε, δύο αιτήματα catch the eye. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λεπτά μόνο. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Μοργάνο ε, για την ε, γνωμοδότησή του και να τονίσω πόσο σημαντικό είναι για μας το θέμα αυτό. Ιδιαίτερα θα ήθελα να εκφράσω την έκπληξή μου για τη θέση αυτή που γενικά συγκρούεται με τη θέση της ΓΚΟΕ. είναι κάτι πολύ θετικό για την Ευρώπη. Θα πρέπει να φροντίσουμε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, ε, όχι μόνο ανάλογα με ε, την απόδοση στα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά και ανάλογα με την διαθεσιμότητα ιδίων πόρων. Τέτοια προσέγγιση χρειαζόμαστε για το μέλλον της Ένωσης. Θα πρέπει να φροντίσουμε η Ένωση να έχει ίδιους πόρους και όχι μόνο κάθε κράτος ε, να συμβάλλει ανάλογα με τη δυνατότητά του, αλλά να έχουμε και έναν προπολογισμό που να βασίζεται στις ευρωπαϊκούς πόρους και όχι μόνο σε εθνικούς. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό πολύ με εκπλήσει η θέση της ΚΟΕ. Το μόνο που θα ήθελα να πω στον κύριο Μοργάνο είναι το εξή. Καταρχά ε, χρειάζεται να να λάβουμε υπόψη μας και το έγγραφο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα μελλοντικά σενάρια για τη χρηματοδότηση της Ένωσης, διότι το έγγραφο αυτό περιέχει όλα τα διαφορετικά σενάρια για νέους τρόπους χρηματοδότησης. Και δεύτερον, θα πρέπει να προσέξουμε το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει νέε προκλήσει όπω είναι ο κοινωνικό πυλώνα, η μετανάστευση, η άμυνα όλα αυτά σημαίνουν ότι θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες. Και τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούν και άλλα θέματα, όπως είναι η τελωνιακή δασμή. Πάντως, γενικά θα στηρίξουμε τη δουλειά του κυρίου Μοργάνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ άκουσα τη συζήτηση. Καταρχά, χαίρομαι ιδιαίτερα για την άποψη του εισηγητή μα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμω, γιατί πρόκειται για μία γνωμοδότηση για το κομμάτι των ιδίων πόρων ε, της Επιτροπής ε, ε, Νομισματικών και δεν αφορά όλες τις δαπάνες. Ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με την πολιτική συνοχή, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει θέση στην έκθεση αυτή. Γι' αυτό Ήθελα να ε, τονίσω ότι το θέμα της φορολογίας πρέπει να τονιστεί όλος ιδιαίτερος γιατί αυτό είναι το βασικό στοιχείο της αρμοδιότητάς μας και πρέπει να το τονίσουμε όσον αφορά τώρα την Ευρωζώνη ε, και πάλι εγώ δεν νομίζω ότι με την ευκαιρία αυτή της γνωμοδότησης που πρέπει να ξαναρχίσουμε ολόκληρη τη συζήτηση για το ε, νομισματικό ταμείο κλπ. γιατί τότε ε, θα δίναμε την εντύπωση ότι ε, συνδέονται οι δύο συζητήσεις. Δεν είναι όμως αυτός ο στόχος της νομοδότησής μας. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια αναφορά προς υπόμνηση, ε, δηλαδή ότι εντάξει περιμένουμε να δούμε τι, αποφάσεις θα τι προτάσεις θα υπάρξουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εγκριθούν από τους συνομοθέτες είτε για το ESM είτε για τον καθορισμό ενός προϋπολογισμού της Ευρωζώνης τότε οι αποφάσεις μας θα προσαρμοστούν. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να συμπεριλάβουμε όλες μας τις θέσεις αυτή τη στιγμή σε αυτήν την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις ε, ε παρεμβάσεις. Ε, Πράγματι, πρέπει να υποβάλουμε ένα, μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Προπολογισμών. Εμείς δεν ορίζουμε το πλαίσιο, αλλά είναι νομίζω πολύ σημαντικό να επαναλάβουμε κάποια στοιχεία επί των οποίων συμφωνούμε, όπως η ενίσχυση της συνοχής, όπως ε, βεβαίως ε, η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. Και θα προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη μας τα θέματα που έθεσαν οι συνάδελφοι που πήραν το λόγο θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε το πόσο είναι εφικτές οι προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα και από την Επιτροπή Μόντι και από τον πρόεδρο Δράγκη. Νομίζω ότι το πρόβλημα το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι να προσπαθήσουμε να δείξουμε τι θέλουμε να κάνουμε με τους ιδίους πόρους Προσωπικά πιστεύω ότι ο κοινωνικός πυλώνας, ο οποίος ε, τέθηκε από συναδέλφους, δημιουργεί κάποιες ανησυχίες οι οποίες είναι σαφείς και πάνω σε αυτές το Κοινοβούλιο έχει εκφραστεί με ξεκάθαρο τρόπο. Δεν έχουμε πια χρόνο στη διάθεσή μας, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Να πω ότι Βλέποντας και το πλαίσιο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη τις τροπολογίες έτσι ώστε να κάνουμε μία πρόταση η οποία να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτική γίνεται. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις έτσι ώστε νομίζω να επιδιώξουμε τις κατευθύνσεις τις οποίες όλοι έχουμε εκφράσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 7η Δεκεμβρίου. Η εξέταση των τροπολογιών 24 Ιανουαρίου και ψηφοφορία ταυτόχρονα. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Σας ευχαριστώ. Τέλος. Θα συνεχίσουμε αύριο. Session 8.15 uh, with Libe Committee. Έχουμε στις 8 και 4 κοινή συνάντηση με τη Λίμπε, με την Επιτροπή Λίμπε.